Dear colleagues, please. Let's start. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε παρακαλώ. Έχουμε την έκτακτη συνεδρίασή μας και ας ξεκινήσουμε καταρχήν με την υιοθέτηση, με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Νοεμβρίου. Εγκρίνονται και τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Και περνάμε στα σημεία 4 και 5. Δύο εκθέσεις που θα τις εξετάσουμε μαζί. είναι τμήμα της μεγάλης δέσμης ε, μέτρων σχετικά με τις τράπεζες. Αποφασίσαμε σήμερα να γίνει η παρουσίαση των τεσσάρων εκθέσεων του κυρίου Χακμάκ ε, και του ε, κυρίου Σάιμον Πίτες και ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές για τις προσπαθίες τους. Ξεκινάμε με ένα πολύ καλό κείμενο από πλευράς Κοινοβουλίου που θα αποτελέσει βάση για συζητήσεις και ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε με την απαραίτητη επιμέλεια και την απαραίτητη ταχύτητα. ώστε να έχουμε ένα καλό ρυθμό στις εργασίες μας και να είμαστε έτοιμοι για τις συζητήσεις με το Συμβούλιο που επίσης προχωρεί με τις ε, εργασίες του για, αυτό, αυτή την υποδέσμη μέτρων, αν μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι. Έχουμε τις δύο εκθέσεις του Γκούναρ Χόκμαν και δίνω το λόγο στον Γκούνερ Χόκμαν για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και αποδεκτών υποχρεώσεων μεταξύ άλλων. Ο κύριος Χόικμαρκ, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους εσάς που, που συνεισφέρετε στην έκθεση αυτή μέχρι τώρα. Δύο σημεία θέλω να αναφέρω που τα θεωρώ πιο σημαντικά από όλα τα υπόλοιπα που συζητούσαμε και που ήταν και πολύ σημαντικά κατά τη σύνταξη της έκθεσης αυτής. Πρώτον, ότι χρειαζόμαστε σταθερές και δυναμικές τράπεζες. Δηλαδή πρέπει να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνεται κατά τρόπον ώστε να υποστηρίζουμε τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Διαφορετικά θα μπούμε σε ένα νέο κύκλο οικονομικής αστάθειας με απώλεια επενδύσεων και απώλεια ανάπτυξης Άρα πρέπει να προχωρήσουμε παράλληλα σε αυτά τα δύο που προανέφερα. Και ως ε, πρώην εισηγητής της VRD ε, θέλω να πω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε δύο σημαντικές πτυχές της οδηγίας για την ε, ανάκαμψη και εξυγένση των τραπεζών. Όταν έχουμε τράπεζες σε αφαιρεγγιότητα, πρέπει να έχουμε ένα τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε και δεν θα πρέπει οι φορολογούμενοι να πληρώνουν τα χρήματα για αυτή την εξυγίανση, αν δεν είναι αυτό απαραίτητο. Αυτά σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, βλέπω ότι χαμογελάτε θετικά για την αναβίωση του καπιταλισμού. Ένα επιχείρημα που θα κερδίσει. Και το δεύτερο σημείο είναι να διατηρήσουμε πειθαρχία στην αγορά, όπως προκύπτει από την οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγένση των τραπεζών. Δηλαδή, όχι μόνο μέσα όπως η διάσωση με ίδια μέσα θα διασφαλίσουν την ε, εξυγένση των τραπεζών, αλλά θα διασφαλίσουμε ότι θα το γνωρίζουν όλοι όταν επενδύουν σε μία τράπεζα εκτίθεται σε κίνδυνο. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που προκύπτουν από την, ανάκαμψη, από την οδηγία για την ανάκαμψη και εξηγένση των πιστοτικών ιδρυμάτων μακροπρόθεσμα, γιατί χρειάζεται μια μακρά διαδικασία μάθηση για να το καταλάβουμε και χρειάζεται κάποιο χρόνο. Αν δούμε τις ε, δύσκολε συνθήκε τα τελευταία χρόνια για τι τράπεζε, είναι σαφέ ότι ακριβώ αυτό είναι το σημείο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά τα προβλήματα για τις τράπεζες και οι αρμόδιες αρχές αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουν. Είναι επίσης ε, σημαντικό για αυτά τα οποία προτείνουμε σε αυτήν την έκθεση η συνολική ικανότητα απορρόφησης ε, ζημιών. Ε, δεν το κάνουμε μόνο για να μιλάμε για το τι συμβαίνει με τη διάσωση με ίδια μέσα. Σημαντικό είναι να πούμε ότι όλα τα κεφάλαια των τραπεζών είναι διασώσιμα με ίδια μέσα αν δεν εξαιρούνται από συγκεκριμένους νόμους και κανονισμούς. Να υπάρχει δηλαδή σαφήνεια και ένα σαφές μήνυμα προς τις αγορές. Όταν λοιπόν μιλάμε για τη συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε δυναμικές και σταθερές τράπεζες, και δεν θέλουμε να θίγονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με επιπλέον υποχρεώσεις για να τηρήσουν τις ελάχιστες απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων και αποδεκτών υποχρεώσεων. Δηλαδή, αν έχουν υψηλό επίπεδο ιδίων κεφαλαίων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να μην αποτελεί πρόβλημα και να χρειάζεται ακόμη υψηλότερε ελάχιστε απαιτήσει, γιατί δίνουμε αντικίνητρα, δίνουμε λάθος κίνητρα στις εταιρείε με χαμηλό επίπεδο κεφαλαίων. Είναι για αυτές εμπόδιο στην αύξηση κεφαλαίων. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου για να υποστηρίξουμε τη σταθερότητα. Τράπεζες που έχουν υψηλότερο επίπεδο κεφαλαίων από ό,τι απαιτεί ο κανονισμός, να το λάβουμε υπόψη για αυτές. Και επίσης εισάγουμε μία ε, ρήτρα ε, διαφύλαξης ε, των κεκτημένων ώστε να λάβουμε υπόψη αυτούς που έχουν τηρήσει την νομοθεσία σχετικά με τις υποχρεώσεις τους. Και τα κεφάλαια μειωμένης εξασφάλισης δεν θα είναι μεγαλύτερο από τις απαιτήσει της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε ελάχιστες απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων και αυτές θα τις ορίζουν οι αρμόδιες αρχές, αλλά το επίπεδο της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών, το, το συγγνώμη, διορθώνει ο το επίπεδο κεφαλαίου μειωμένη εξασφάλισης δεν θα είναι υψηλότερο από το TILAC, τη συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών. Πολλές συζητήσεις έγιναν για το επίπεδο του MRL. Προτάθηκαν από 5 έως 2 ημέρες μορατόριου και αυτό συζητήθηκε πολύ και θα ήθελα να σας εξηγήσω γιατί. Πρώτον, αν βάλετε ένα ίδρυμα, ένα πιστοτικό ίδρυμα σε μορατόριου, σε δυνατότητα αναστολής των υποχρεώσεων πληρωμής, αυτό είναι ένα μήνυμα του ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει και αν αυτό το μορατόριου συνεχίζεται, όσο περισσότερο συνεχιστεί, τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα αξιοπιστίας θα έχει. Και για να το πω πιο απλά, αν οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να αξιολογήσουν το πρόβλημα σε δύο μέρες, η αγορά θα πει άρα υπάρχει πρόβλημα. Και στην πραγματικότητα η τράπεζα έχει, θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Άκουσα το επιχείρημα ότι χρειάζονται περισσότερε μέρε από δύο και καταλαβαίνω και αυτά τα επιχειρήματα. Εμεί τι ακριβώ κάναμε. Εμεί εφαρμόσαμε την οδηγία BRD που δίνει ένα σαφή οδικό χάρτη για την εξήγηση των τραπεζών Δεύτερον, πρόσφατα εγκρίναμε νομοθεσία για την ιεράρχηση που μας δίνει ένα σύντομο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των τραπεζών και στην οδηγία ανάκαμψη και εξυγίανση έχουμε και μια απέτηση για το σχέδιο εξυγίανση, δηλαδή ένα οδικό χάρτη για το τι πρέπει να γίνει για την εξυγίανση. Και τώρα βάζουμε και τι διατάξει για τα κεφάλαια μειωμένη εξασφάλιση μέσω του TILAC. δεν προσπαθούμε να κάνουμε πιο δύσκολη την αξιολόγηση των σημαντικών προβλημάτων των τραπεζών, αλλά δίνουμε στις αρμόδιες αρχές ε, ξεκάθαρα εργαλεία για το πώς να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε συζήτηση, γιατί δεν είναι επιστημονικά τα κριτήρια να πούμε ότι δύο μέρες πρέπει να είναι το μορατόριο και όχι παραπάνω, αλλά πρέπει να προσέχουμε αν θέλουμε να επεκτείνουμε το χρόνο για το μορατόριο, γιατί όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος, τόσο μεγαλύτερο θα είναι ο κίνδυνος η εγχείρηση να επιτύχει και ο ασθενής να αποθάνει. Και θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα fast track, μια ταχεία διαδικασία όταν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αυτά από τις αρμόδιες αρχές. Με την πρότασή μου λοιπόν κύριε Πρόεδρε προσπαθώ να παρουσιάσω το TLAC με τρόπο ώστε να μην θέτουμε σε κίνδυνο τα καλά στοιχεία της BRRD διασφαλίζουμε τη σταθερότητα φροντίζοντας να είναι και δυναμικές οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και διασφαλίζουμε ότι υπάρχει ένα σαφής οδικός χάρτης για όλες τις αρμόδιες αρχές και αυτό γίνεται και με την ταχεία διαδικασία που ήδη έχουμε για την ιεράρχηση. Το πρώτο τρίτο λοιπόν του πακέτου των μέτρων το έχουμε ολοκληρώσει και Ευχαρίστω θα ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων και θα κάνουμε τι συζητήσει με του χιώδει συζητητέ και όποιον άλλον ενδιαφέρεται. Θέλω να καταλήξουμε σε ισχυρή νομοθεσία και στα δύο αυτά στις δύο νομοθετικές προτάσεις και να προσθέσω και κάτι προσβλέπω με χαρά στη συνεργασία με τον κύριο Σίμαν. Και ο κύριος Πίτερ Σέιμον το ίδιο φαντάζομαι, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την εξαιρετική παρουσίασή σας. Να ακούσουμε τους κοιόδης συζητητές. Ο κύριος Σίλβε Περέιρα πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη που καθυστέρησα γιατί ήμουν σε μια άλλη συνεδρίαση. Βεβαίως και ξέρουμε περί την πρόκειται. Μιλάμε για την αναθεώρηση τις οδηγίες για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση των Τραπεζών και τον κανονισμό για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Η δική μου αξιολόγηση είναι ότι το γενικό πλαίσιο της BRD παραμένει ορθό. Ο κύριος στόχος αυτής της αναθεώρησης είναι να συμπεριλάβουμε και τα διεθνή πρότυπα TILAC για τη συνολική ικανότητα απορρόφησης ε, ζημιών να τα ενσωματώσουμε στην υφιστάμενη, στις υφιστάμενες απαιτήσεις ε, MRL. Έχει σημασία αυτή τη στιγμή για την Επιτροπή η εφαρμογή του άρθρου 55 για την αναγνώριση της διάσωσης με ίδια μέσα. Και καταρχήν εγώ θέλω να χαιρετήσω το προτινόμενο πακέτο μέτρων από την Επιτροπή. Γενικά μας ικανοποιεί η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν και πρέπει να γίνουν κάποιες σημαντικές βελτιώσεις. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Χόκμαρκ, για αυτό το σχέδιο έκθεσης, που αποτελεί μια καλή βάση για να συνεχίσουμε την δουλειά μας. Εδώ κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων, οπότε έχω κάποιες προκατακτικές παρατηρήσεις. Δύο σημεία θεωρώ πολύ σημαντικά για την αναθεώρηση αυτή. Το πρώτο είναι η βαθμονόμηση των ελάχιστων απαιτήσεων, των MRL, και το θέμα των μεταβατικών διατάξεων για το MRL. Η βαθμονόμηση των ελάχιστων απαιτήσεων MRL πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένη, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα εξηγήσεων των τραπεζών σε υψηλότερο επίπεδο και να ενισχυθεί και η οικονομική σταθερότητα. Αλλά παράλληλα οι τράπεζες θα πρέπει να παραμένουν σε θέση να χρηματοδοτούν την οικονομία. Και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό οι απαιτήσει MRL να μην είναι υπερβολικά βαθμονομημένες και να μην απαιτείται από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να τηρούν ελάχιστες απαιτήσει MRL δυσανάλογες προς τις ανάγκες εξυγένσής τους. Περαιτέρω, σχετικά με την βαθμονόμηση MRL, βλέπω ότι η τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής ε, Αρχής Τραπεζών για το MRL διαπιστώνει ότι θα είναι δύσκολο να τηρηθούν οι απαιτήσεις MRL και αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε, διότι είναι σοβαρό όταν κάνουμε τη βαθμονόμηση των απαιτήσεων MRL. Τώρα για τη μεταβατική περίοδο για τις απαιτήσει MRL θα πρέπει να έχουμε με τέτοια μεταβατική περίοδο, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να γίνει σταδιακά η εισαγωγή των απαιτήσεων MRL, γιατί μπορεί οι αγορές να δυσκολευθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να εξασφαλίσουν μεγάλα κονδύλια. Χρειάζεται μια εναρμονισμένη ελάχιστη περίοδος για συμμόρφωση με τα MRL και για κάποια ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορεί να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια σε κάποιες περιπτώσεις. Η πρόταση της Επιτροπής για δύο νέα εργαλεία που ανέφερε ο κύριος Χόκμαρ και το Μορατόριου ε, ε, ένα μορατόριο μου πέντε ημερών μπορεί να δημιουργεί ανησυχίε. Μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό το να έχουμε πέντε μέρες. Μπορεί να υπονομεύει την εμπιστοσύνη, να οδηγήσει ακόμη και ε, σε bank run και να ε, υπονομεύσει τη θέση των τραπεζών. Έχουμε δύο και δύο νέα εργαλεία με δύο ημέρες το καθένα και αυτό ίσως είναι πιο λογικό, αλλά θα πρέπει να επανέλθουμε σε μελλοντικές συζητήσεις στα θέματα αυτά. Τώρα όσον αφορά τις αποδεκτές υποχρεώσεις του MRL δεν θα πρέπει να προχωρούν πέραν του προτύπου ΛΑΚ. Και εδώ συμφωνώ με τον εισηγητή. Επίσης συμφωνώ με τον εισηγητή σχετικά με το θέμα της ε, ρήτρα ε, προστασίας και εκτιμένων δικαιωμάτων. Πρέπει να επιτρέψουμε μια τέτοια ρήτρα για τα ε, υφιστάμενα χρέη. Όσον αφορά τα κεφάλαια μειωμένης εξασφάλισης, θα πρέπει να ισχύει για τις παγκόσμιες συστημικές τράπεζες και για τα υπόλοιπα ιδρύματα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο. Θα γίνουν πολλές συζητήσεις σχετικά με το MRL στο μέλλον. Δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι θα πρέπει από την BRD να εξαιρούνται οι καταθέσεις δημοσίων φορέων από την διάσωση με ίδια μέσα, διαφορετικά τίθεται σε κίνδυνο χρήματα των φορολογουμένων και αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Η αναθεώρηση αυτής της δέσμης μέτρων σίγουρα θα χρειαστεί πολλές συζητήσει γιατί θα ακουστούν πολλές και διαφορετικές απόψεις, αλλά να μην ξεχνάμε ότι θέλουμε να επιτύχουμε μια εξυγίανση αποτελεσματική διατηρώντας την χρηματοοικονομική σταθερότητα και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας και με τον εισηγητή κατά τους προσεχείς μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Θα σε ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους του ECR. Ο κύριος Φόξ εκ μέρους του κύριου Καμάλ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Καμάλα ε, θα ήθελα να σας δει, συγγνώμη γιατί δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης, το οποίο και καλεσορίζει. Η ομάδα μου στηρίζει τις τροπολογίες για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και αποδεκτών υποχρεώσεων για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, για το grandfathering, για τη μία απαξίωση όλων αυτών ε, των αποθεμάτων κεφαλαίου. Θα πρέπει να υπάρχει grandfathering σε όλα αυτά τα κονδύλια και κεφάλαια. Το μορατόριο μου στις συνθήκες με, το, με τις οποίες προτείνεται παρουσιάζει κάποια θέματα γιατί ε, έχουμε επεκτείνει παραπάνω από το προθεσμία των δύο ημερών και έχουμε πάει στις έξι ημέρες και αυτό θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την οικονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη της αγοράς. Δεν γίνεται αξιολόγηση αντικτύπου για τις αλλαγές αυτές και πολλοί εμπλεκόμενοι μου είπαν ότι αυτό θα επηρεάσει το επίπεδο συμμετοχής τους σε επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι ε, θα εκτίθεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο και δεν θα μπορούν να αποσύρουν τις επενδύσεις τους μετά από εύλογο χρονικό διάστημα. Γιατί λοιπόν να επενδύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ άλλες αγορές τους προσφέρουν αυτή την προθεσμία των δύο ημερών. Εγώ στηρίζω την διεθνώς αποδεκτή προθεσμία των δύο ημερών και ε, οι εθνικές αρχές να μπορούν να την ξεπεράσουν μόνο όταν αυτό απαιτείται υπό κατεπίγουσες και κατεξαίρεσιν συνθήκες. Τώρα, για τις ελάχιστες απο... ε, απαιτήσεις της τροπολογίας 2 και 13 που έχουν να κάνουν με το δεύτερο πυλώνα, έχω να πω ότι δεν υπάρχει καθόλου ευελιξία και ούτε περιθώριο ελιγμών για τις εθνικές αρχές και δεν μπορούν να καθορίσουν το επίπεδο των μειωμένης εξασφάλισης ε, χρεών και τη στρατηγική για την αντιμετώπιση όλων αυτών. Νομίζω ότι οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών τηρώντας πάντοτε την αρχή της αναλογικότητας. Στηρίζω την αρχή της αναλογικότητας που διέπει την πρόταση του εισηγητή. Πράγματι, οι μικρές τράπεζες δεν μπορούν να ε, ανταπεξέλθουν στις ίδιες προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα όπως οι μεγάλες και έχει δηλωθεί ότι οι απαιτήσει για τις μικρότερες τράπεζες ήταν υπερβολικές, δυσανάλογες και ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει μέρος της διατύπωσης του κείμενου. Η ομάδα μου έχει κάποιες επιφυλάξεις για το guidance, για τις οδηγίες για το MRL, για τις ελάχιστες απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων και αποδεκτών υποχρεώσεων. Εμείς είμαστε υπέρ της διαγραφής του guidance και με ενδιαφέρον θα ακούσω και τις απόψεις των συναδέλφων για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ, Κορνίγια, για εξ των Φιλελεύθερων. Ευχαριστώ. Α, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω δύο λόγια εκ μέρου του συναδέλφου κυρίου Κορνίγε που δεν είναι εδώ σήμερα. Θέλει να ευχαριστήσει τον κύριο Χάκμαρκ για αυτό το πολύ καλό σχέδιο έκθεση, το οποίο ε, κομίζει σημαντικέ διευκρινήσει. Το γεγονό ότι η αρχή εξυγίανση θα ασχοληθεί αναπερίπτωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και με, ε, και με το TILAC, όλα αυτά είναι πολύ καλά. Και όλα αυτά απεικονίζουν και απηχούν τις επιθυμίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί πολύ συχνά οι ε, στελέχοι της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας έχουν τονίσει πόσο σημαντική είναι η αλλαγή της βαθμονόμησης όλων αυτών των ελάχιστων απαιτήσεων. Έχω κάποια ερωτηματικά να θέσω. Ποια είναι η πραγματικότητα ως προς τα MRL εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλουμε τραπεζική ένωση, τότε πρέπει να τη θεωρούμε ως χώρο ενιαίας και μοναδικής δικαιοδοσίας. Να έχουμε μία και μόνη ελάχιστη απέτηση και όχι πολλές και διαφορετικές ελάχιστες απαιτήσει εντός ε, του ιδίου όμιλου ή της ίδιας ομάδας είναι αυτός ο, ο μηχανισμός, ο μοναδικός μηχανισμός ε, τραπεζών. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ε, τροπολογία 20 και διότι το περιεχόμενο της συμβάλλει στο κατακαιρματισμό της εποπτείας και της διαδικασίας εξυγίανσης. Θα πρέπει η διαδικασία εξυγίανσης του ομίλου να είναι διαυγής και να μην είναι όμοιροι όλοι μεταξύ των χωρών προέλευσης και χωρών υποδοχής. Και τέλος, ως προς το μορατόριο, ο εισηγητής φέρνει κάποιες διευκρινήσεις πολύ ευπρόσδεκτες, ωστόσο δεν ξέρω αν ε, διευκρινίζει την κατάσταση ε, περισσότερο. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν σε θέση να μας διαφωτίσει. Ευχαριστώ για τους πράσινους. Όχι, συγγνώμη. Για την ΚΟΕΠ. Ο κύριος Σούντερβεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και κυρίως ευχαριστώ τον εισηγητή και αποφελούμε της ευκαιρίας να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων που και εκείνος ξεκίνησε με κάποια πολιτικά επιχειρήματα. Δεν ξέρω αν θα αναβιώσουμε τον καπιταλισμό γιατί ως εκπρόσωποι της αριστεράς δεν νομίζω ότι αυτή είναι η πρόθεσή μας. Πιστεύω ότι η έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας μας δίνει τη δυνατότητα ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών να φροντίσουμε τις λεπτομέρειες για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη σταθερότητα για τις τράπεζες. Και μου φαίνεται ότι σε πολλά σημεία υπάρχουν θετικά σημεία, διότι φαίνεται ότι έχουμε λάβει υπόψη τα διδάγματα από την ε, χρηματοοικονομική κρίση πριν από λίγα χρόνια. Και ίσως είναι επιχειρήματα αυτά τα οποία πρέπει να δυναμωθούν. Και νομίζω ότι και ο κύριος Ντάισελμπλουμ στο Eurogroup ε, είχε διαπιστώσει ότι σε σχέση με τη διάσωση της ε, Ελλάδας κατά την ελληνική κρίση είχαν διαπραχθεί σφάλματα και ίσως το, η ανάγκη μεγάλης διάσωσης ε, ήταν ένα βασικό σφάλμα. Τώρα προσπαθούμε να έχουμε διάσωση με ίδια μέσα για να αντιμετωπίσουμε ε, θέματα θερεγγιότητας τραπεζών χωρίς ε, να επιβαρύνονται μόνο οι φορολογούμενοι στο μέλλον. Η έκθεση προς το παρόν ε, δεν νομίζω ότι πλήρει όλες τις προϋποθέσεις που θα θέταμε ε, για μια ικανοποιητική έκθεση. Τα μέσα αυτά τα οποία παρουσιάσατε, το TILAC και το MRL, δεν νομίζω ότι λειτουργούν κατά τον τρόπο που παρουσιάσατε από την πλευρά της αριστερής πτέρυγας. Νομίζω ότι ε, προσπαθούν ε, να ενισχύσουν ε, τις συστημικές τράπεζες. Στο μέλλον θα έχουμε την ευκαιρία για επικοδομητικές συζητήσεις για να μπορέσουμε να ε, συζητήσουμε και τα πολιτικά ζητήματα αλλά και τις τεχνικές και διοικητικές τροποποίησεις που μπορεί να χρειαστούν. Στις τροπολογίες που θα υποβάλουμε θα κάνουμε μια σειρά προτάσεων για βελτίωση του κειμένου για να βελτιώσουμε την ασφάλεια δικαίου ούτως ώστε να είναι δυνατή η διάσωση με ίδια μέσα και να μην επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι. Για τη βαθμονόμηση των απαιτήσεων MRL που ήδη αναφέρθηκε φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε σε διάσωση και πάλι και σε θέματα που αφορούν το άρθρο 55 και την διάσωση υπό τη μορφή του bail-out. Κάποιες τροπολογίες που προτείνατε για την μείωση των αρμοδιοτήτων των ε, αρμοδίων αρχών ε, δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Οι απαιτήσει MRL δεν θα πρέπει να ε, υπερβαίνουν τα επίπεδα του προτύπου TILAC. Ένα άλλο σημείο που αναφέρθηκε επίσης και που θα πρέπει να τονίσουμε αφορά την καθοδήγηση σε σχέση με το MRL. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι παραβιάσεις θα πρέπει και να τιμωρούνται. Όσον αφορά την προληπτική κεφαλαιοποίηση, φαίνεται σαν να πρόκειται για ε, ένα στην πράξη opt-out από την ε, δυνατότητα διάσωσης με ίδια μέσα. Αυτό το οποίο θα θέλαμε να αποφύγουμε δηλαδή. Στο άρθρο 55, στην παράγραφο 2 συγκεκριμένα, Θέλω να πω ότι για μας ε, η διατάξεις του άρθρου 55 σχετικά με τη δυνατότητα διάσωσης ε, με ίδια μέσα είναι πάρα πολύ σημαντικές και στο άρθρο 2 διατυπώνονται ε, εξαιρέσεις και θα πρέπει να δούμε για ποια πιστοτικά ιδρύματα μπορούν να ισχύσουν αυτές οι εξαιρέσεις και μετά τον κύριο Ντάξερπλουν θα μπορούσα να αναφέρω και τον κύριο Σόιμπλε που μίλησε για μείωση ε, των ε, ε, μέσων που επιφέρουν κινδύνους στην κρίση των τραπεζών. Και εμείς ως ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς με τις τροπολογίες μας θα φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε προστασία για τους ε, ε, φορολογουμένους και αυτό θα γίνεται και προς όφελος ε, του ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας ασφάλεια δικαίου και όπως είπαμε από την αρχή θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για τους πράσινους τώρα. Έρνες Ορτασούν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για τις προτάσεις αυτές. Με ενδιαφέρον θα συνεργαστούμε στις συνεδριάσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Καλωσορίζουμε τη θέσπιση του TILAC στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και της BRD Καλωσορίζουμε τη θέσπιση διαφόρων παρατηρήσεων από τον εισηγητή. Συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με το στοιχείο της αναλογικότητας. Προτεραιότητα για την ομάδα μας είναι η ισορροπία μεταξύ της δημιουργίας του κινδύνου και του μοιράσματο του κινδύνου. Με αυτό το φάκελο θα πρέπει να μειωθούν σημαντικά οι κίνδυνοι για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Η θέση του εισηγητή ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νέα στοιχεία που εισάγει ο εισηγητής δεν μας πείθει αυτή η πρόταση μείωσης ε, της περίοδου του μορατόριου από πέντε μέρες σε δύο. Είναι απαραίτητο να έχουμε περισσότερο χρόνο για να εφαρμόσουμε τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης και θα πρέπει να ε, εξαιρεθούν και οι καταθέσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το μορατόριο. Ε, αυτή είναι και μία από τις προτάσεις μας. Το την τροπολογία 16 και το περιεχόμενό της ε, πρέπει να είναι δείκτης αναφοράς για την αξιολόγηση και όχι προαπαιτούμενο. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο και να έχουμε αποφυγή σύγκρουση συμφερόντων, παρακολούθηση από κάλυψη μέτρων, βοήθεια από μη επαγγελματίε και επαγγελματίε επενδυτέ συμβούλου και ούτω καθεξή. Σημαντικό είναι να αντλήσουμε τα διδάγματα από τις πρόσφατες εμπειρίες που είχαμε από την εφαρμογή για την, της για την ανάκτηση και εξυγίανση των τραπεζών, τις εμπειρίες με τον Banco Popular αλλά και διάφορες Ιταλικές τράπεζες. Στο Banco Popular, στην Ισπανική αυτή τράπεζα, δεν υπήρχε αυτή η λίστα με το bail-in εκεί που τη χρειαζόμασταν. Και πρέπει να τροποποιήσουμε το άρθρο 10 έτσι ώστε αυτή η καταγραφή να είναι μέρος του σχεδίου εξυγίανσης και η εκδοχή ενημερωμένη θα πρέπει να διατίθεται εντός 24 ε, ωρών και θα πρέπει να ενημερωθούν τα άρθρα 14, 15, 16 έτσι ώστε ε, να καταστεί σαφές ότι αν κάποια τράπεζα δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτό το προεπαιτούμενο τότε δεν μπορεί να προχωρήσει με τη διαδικασία εξυγίασης. Ως προς αυτή την οδηγία για την ανακτήση και εξυγίαση τραπεζών πρέπει όλα αυτά τα σχέδια να ενημερώνονται και να έχουν καταχωριστεί και να είναι ξεκάθαρα. Μπορεί λοιπόν να βελτιωθεί η διατύπωση στο άρθρο 6 και 7 για την ανάκτηση, recovery, bank recovery και να ε, ενώ το, μπορεί να τροποποιηθεί και το άρθρο 27 για να έχουμε σαφές χρονοδιάγραμμα για την πυροδότηση των μέτρων έγκαιρης παρέμβασης εάν η εβδομαδιαία παρακολούθηση των δικτών δείχνει ότι οι ελάχιστες απαιτήσει ίδιων κεφαλαίων και αποδεκτών υποχρεώσεων και στην οδηγία για την ανάκτηση και εξυγίαση τραπεζών αλλά και στο σχετικό κανονισμό για τις απαιτήσει για τα ίδια κεφάλαια δεν πληρούνται. Αυτά είναι τα μήνυμα, τα ελάχιστα που μπορούμε να διδαχθούμε από την περίπτωση του Banco Popular. Όταν τα κριτήρια δεν πληρούνται, εκεί θα υποβάλουμε τροπολογίες για το άρθρο 32 και κάτι που ανησυχεί την ομάδα μας ιδιαιτέρως είναι το κριτήριο του δημοσίου συμφέροντος έτσι όπως το αξιολογούν ή δεν το αξιολογούν οι αρχές. Έχουμε δει σε ορισμένες περιπτώσεις ότι η αξιολόγηση των αρχών δεν συμπεριέλαβε τα χρήματα του φερολογωμένου όταν εφάρμοσε τα θέματα της αφαιραγκαιότητας στην εθνική νομοθεσία. Πώς αξιολογούμε λοιπόν το δημόσιο συμφέρον. Θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν αυτά τα κριτήρια. Από εκεί και πέρα, παραδοσιακά η ομάδα μας ανησυχεί ιδιαίτερος για την κατάχρηση της προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και βεβαίως θα περιμένετε από εμάς τροπολογίες για να αφαιρεθεί αυτό το εργαλείο. Και για το, ε, τις ελάχιστες απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων και αποδεκτών υποχρεώσεων και για το ΤΙΛΑΚ, για τη συναλλική ικανότητα απορρόφησης ζημιών, εμείς ε, θεωρούμε ότι πρέπει να προσθεθεί στο κείμενο το minimum rational, μια ελάχιστη δηλαδή συλλογιστική, να προσθεθεί η λέξη at least, τουλάχιστον. Ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων θα, για τα G-Funds πρέπει να επεκταθεί για να συμπεριλάβει και το OS2, δηλαδή τα ιδρύματα που είναι σημαντικά για το σύστημα, αλλά και τα ιδρύματα τα χρηματοπιστωτικά που είναι σημαντικά παγκοσμίω για το σύστημα, ε, OS2 και GS3. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά αυτομάτως θα πρέπει να καθίστανται απαιτητά, να υπάρχει να θεωρούνται προαπαιτούμενα, ή αλλιώ να μην μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία εξυγίανσης. Και είναι πολύ σημαντικό επόδιο για την εξυγίανση μιας τράπεζας όταν δεν εκπληρώνει τα κριτήρια για, το TILAC, τη συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών. Σε κάθε περίπτωση είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε επικοδομητικά για να βρούμε λύσεις σε όλα τα εκκρεμή ζητήματα. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι υπάρχει πολλή δουλειά. Είναι σημαντικό να σας υπενθυμίσω ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για την ανάκτηση και εξηγένση των τραπεζών θα γίνει του χρόνου. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά επιτρέπετε να τα θίγουμε αυτά τα ζητήματα, έτσι δεν είναι μια ερώτηση να κάνω, απλά, λέει ο κύριος Ορτασούν. Ναι, βεβαίως, λέει ο Πρόεδρος. Γιατί θα ήταν καινούριο και νέο ε, ο πρόεδρος να περιορίσει τις ικανότητες και τις δυνατότητες των μελών της ομάδας. Ο πρόεδρος, όχι, απλά έλεγα ότι είναι ενδιαφέρον να μείνει κανείς στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου κειμένου, αλλά δεν πρόκειται να απορρίψω τις τροπολογίες. Ο φάκελος για τις ελάχιστες απαιτήσει ίδιων κεφαλαίων και αποδεκτών υποχρεώσεων δεν είναι ίδιος με την οδηγία για την ανάκτηση και εξυγίανση τραπεζών που θα αναθεωρηθεί του χρόνου με την πρόταση της Επιτροπής. Επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Κύριε Βουά, ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαίρω και εγώ τον εισηγητή. Σύντομα συζητάμε για αυτά τα κύρια σημεία και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε. Ως πρώτο κύριο σημείο να πω και λυπάμαι που το υπενθυμίζω γιατί είχαμε την έκθεση δική σας όπου ήσασταν εσείς για την αναθεώρηση των τραπεζών που τελικά το καταλήψαμε ώστε να προστατεύσουμε τους αποταμιευτές και τους καταθέτες γιατί χωρίς εκείνη την νομοθεσία το Μπέιλιν στην ουσία γίνεται μάταιο. Το γεγονό λοιπόν ότι η Κομισιόν αποφάσισε διαφορετικά οδήγησε όλο το πακέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάζει κάποια κενά και τον επόμενο κύκλο συζητήσεων. Δυστυχώ θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό το κενό όσον αφορά την αναδιάρθρωση των τραπεζών και μεταρρύθμιση του συστήματο λειτουργία. Για το μορατόριο μου έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση στην Ιταλία και νομίζω η κατεύθυνση του εισηγητή είναι σωστή γιατί πρέπει βεβαίω οπωσδήποτε να μειώσουμε απολύτω τον χρόνο κατά του οποίου μπλοκάρονται οι καταθέσεις έστω και για μια μέρα, για μια ώρα, ένα μπλοκάσμα αυτών των χρημάτων θα δημιουργούσε πανικό στους αποταμιευτές και θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στην τράπεζα και στο τραπεζικό σύστημα που αφορά την εξηγία της τράπεζας. Γι' αυτό λοιπόν είμαι αντίθετος. Θα πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Θεωρώ ότι επειδή εδώ θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό πανικού που θα πρέπει να αποφύγουμε. Εξάλλου νομίζω ότι οι αρχές εξυγίανσης δεν έχουν κανένα δικαίωμα να μπλοκάρουν τους ε, λογαριασμούς των καταθετών και να μην μπορούν οι κάτοχοι λογαριασμού να κάνουν αναλήψεις από το λογαριασμό τους. Πρέπει λοιπόν να είναι ενημερωμένοι πρώτα οι καταθέτες και μετά να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Μετά έχουμε και κάποιες ανησυχίες σε σχέση με τους επενδυτές και τα εργαλεία τα οποία αφορούν το χρέος πριν από την ημερομηνία ορίμανσης. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να θεσπίσουμε εξαιρέσεις για το bail-in όσον αφορά τους μικροκαταθέτες. Γιατί καταλαβαίνω ε, όταν κάποιος ας πούμε υπογράφει ένα χαρτί αναλαμβάνει τους κινδύνους όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πάρα πολλά άτομα δεν γνωρίζουν ακριβώς τι προϊόντα χρηματοοικονομικά αγοράζουν ιδιαίτερα με όλη αυτή τη ρευστότητα που έχουν διαθέσει οι κεντρικές τράπεζες νομίζω οι αποδόσεις έχουν μυθεί κατά πολύ οπότε πάρα πολύ εύκολα ε, οδηγούμε ε, στην απόγνωση τους μικροπαιδητές. Και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους όταν θα εφαρμοστούν οι νομισματικές πολιτικές. Οι ευθύνε λοιπόν για τους μικρούς δεν θα πρέπει να είναι στις δικές, του τους ώμου και δεν θα πρέπει να έχουν μπροστά του το φόβετρο του Μπέιλιν. Εμείς στην Ιταλία είχαμε την εμπειρία, επειδή, αυτή την εμπειρία αυτή, επειδή δεν ήταν καθόλου θετικό να υπάρχουν άτομα τα οποία στο χαρτοφύλλο του είδαν να ξαναμίζονται οι καταθέσεις τους. Αυτό το είδαμε. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτά τα θέματα. Μετά, όσον αφορά τους μηχανισμούς αποζημίωσης, σε περίπτωση πώλησης προφίλ επενδυτικού όταν δηλαδή έχουμε κατάλληλα εργαλεία και όταν προβλέπεται κάποια αποζημίωση θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης, διαχείρισης αυτού του είδους πρακτικών γιατί υπάρχει βεβαίω η ευθύνη από τις τράπεζες σε αυτές τις περιπτώσεις οπότε οι καταθέτες θα πρέπει να μην αποζημιώνονται τη στιγμή που δεν έχουν και τις αρμοδιότητες αλλά ούτε μάλλον στις αρμοδιότητες ούτε την δυνατότητα να αποτιμήσουν, να αξιολογήσουν το δυναμικό των επενδύσεων που έχουν κάνει. Αυτή ήταν λοιπόν η εμπειρία που είχαμε στην Ιταλία με την εξυγίανση των ε, τραπεζών μας και είδαμε ότι υπήρξαν κάποια σοβαρά προβλήματα. Ίσως να μην τα αντιμετωπίσατε και εσείς σε άλλες χώρες αντίστοιχες καταστάσεις, αλλά εμεί ε, δοκιμάσαμε πραγματικά στο πετσί μας αυτές ακριβώς τις ε, διακασίες, αυτά τα φαινόμενα. Όταν δηλαδή εφαρμόζεται ένας κανόνας, ο οποίος είναι άτεκτος και προκαλεί συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Μόνο, εκ μέρους του Τσάνη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά. Μεταφέρω την άποψη του κυρίου Ζανή αυτές τις δύο εκθέσεις. Ο κύριος ε, Ζανή δεν μπορεί να έρθει για το πρώτο κομμάτι, Θα έρθει όμως το δεύτερο, έκθεση του κ. Σάμαν Πίτερ. Τα περισσότερα μου σχόλια αφορούν το 61 και το 63 κείμενο. BRRD, το άρθρο 45. Η προσπάθεια σύγκλησης υπολογισμού στο ΕΜΡΕΛ σχετίζεται με το TILAC. Θεωρητικά αυτό είναι σωστό, όμως στην πράξη θα έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά τον κίνδυνο και τις αποδόσεις των πολύ μικρών τραπεζών που δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα δικά τους εργαλεία για την αξιολόγηση του κινδύνου. Οπότε η χρήση ε, προτύπων, ενιών προτύπων, δίνει πάντοτε υψηλότερη εκτίμηση του κινδύνου από τα εσωτερικά πρότυπα που έχουν μικρές τραπεζές. Οπότε η στάθμιση αυτών των κινδύνων είναι εις βάρος των μικρών τραπεζών που θα έπρεπε να εκδώσουν σε υψηλότερο κόστος περισσότερα MRL. Και αυτό θα οδηγήσει βεβαίως στην εξαγορά του από μεγαλύτερες τράπεζες και στον περιορισμό των δραστηριοτήτων και σε αναζήτηση κινδύνου. Για 361 που αφορά την εξυγίανση ένα τμήμα των σχολείων ταυτίζεται με το 362 γιατί στην ουσία έχουμε το ίδιο περιεχόμενο με το άρθρο 45 του 362. Το νέο 45β του 362 μας δημιουργεί κάποια σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την προστασία των αποταμιευτών. Δηλαδή, στα πλαίσια του MRL παράγωγα προϊόντα τα οποία έχουν ε, επιπτώσει επίπεδο ε, επιτοκίων, όμως όχι σε επίπεδο κεφαλαίου. Αυτά τα προϊόντα συνήθως ε, πολλούνται στους ιδιώτες καταθέτες. Η δυνατότητα λοιπόν αποζημίωσης είναι σημαντική όσον αφορά την προστασία των επενδυτών αυτών. Το κόστος σε περίπτωση bail-in αποτελεί ένα μεγάλο κίνδυνο και μπορεί να φαίνεται παράξενο να έχουμε έναν Ευρωπαίο νομοθέτη ο οποίος στην ουσία οδηγεί στην ε, απώλεια, σε απώλειες των ε, μικροκαταθετών υπέρ των μεγάλων τραπεζών που διαθέτουν αυτά τα προϊόντα. Τώρα το 361 και το 12β είναι σχεδόν ταυτόσιμο όσον αφορά το περιεχόμενο του 45β στο 362. Έχουμε το 45ε, ε, το οποίο θεσπίζει ε, μια νέα ερμηνεία ε, της BRRD όσον αφορά την εξηγένση. Θεωρούμε ότι ο τρόπος υπολογισμού του MREL ήδη οδηγεί σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητα όσον αφορά τι αρχέ εξυγίαση, που ήδη αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο αστάθεια. Στο 45 λοιπόν ε, εδώ στην ουσία ανοίγουμε το δρόμο για τη δημιουργία επιπλέον Εμρελ σε πλήρη περίοδο κινδύνου όσον αφορά τα λόγω ιδρύματα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι επιθυμητό. Και το 12F του 361 επισύρει τα ίδια σχόλια με το 45 ε του 362. Τέλος, το πιο σημαντικό κατά την άποψή μας είναι οι τροπολογίες στα 27 και 63, όπως και το 29α νέο άρθρο όσον αφορά το μορατόριου, ε, που τα θεωρούμε αυτά τα άρθρα πολύ επικίνδυνα. Το να ε, εφαρμόσουμε ένα πάγωμα των δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα όσον αφορά την, τις αναλήψεις κεφαλαίων, ε, θεωρητικά θα μπορούσε να, να είναι κάτι το θετικό, αλλά στην πράξη, όσον αφορά το μορατόριο μου, δεν θα μπορέσει παρά να οδηγήσει στην πτώση, στην πτώχευση του λόγου Όταν έχουμε ένα πάγωμα μετά την περίοδο των πέντε ημερών, θα έχουμε ε, πλήρη διαρροή κεφαλαίων, διαφυγή κεφαλαίων και θα τρέξει ο κόσμο ω τι αποταμιεύσει του. Επίση, ε, προβλέπουμε ότι δεν θα εφαρμοστεί τον ίδιο τρόπο το πάγωμα θα είναι πλήρες για τους ιδιώτες, αλλά θα το παρακάψουν άλλοι πιο ισχυροί παράγοντες ή φορείς. Συνολικά, Πρόεδρε και κύριε Σιγητά, θεωρώ ότι αυτές οι δύο αναθεωρήσεις που μας προτείνονται, θεωρούμε ότι επιφέρουν περισσότερη αστάθεια και αβεβαιότητα σε ένα ήδη ατελές περιβάλλον Τραπεζικής Ένωσης. Τραπεζική Ένωση που ήδη είχε επιφέρει αστάθειες και αβεβαιότητες όσον αφορά τους επενδυτές. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχει ενισχυθεί ο κίνδυνος και απειλεί τους ε, καταθέτες στις πιο μικρές τράπεζες, τις πιο τοπικές, αυτές που η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή θα ήθελε να εξαφανιστούν όσον αφορά την ύπαρξη της διασυνοριακή τραπεζικής αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία the Eye. Ο κύριος Μπάλτς έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, χαιρετίζω το έργο του Γκουναρ ε, Χέκμαρκ που μαζί με τον Πέτερ Σίμων μας παρουσιάζουν ε, αυτή τη δέσμη μέτρων για τη μείωση των κινδύνων την δέσμη αυτή μέτρων πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία και είναι μια δύσκολη ισορροπία. Από τη μια μεριά θέλουμε να δυναμώσουμε τις τράπεζες, από την άλλη πλευρά να προστατεύσουμε τους φορολογουμένους. Χωρίς να ε, περιπλέξουμε υπερβολικά τις διατάξεις για την εξυγίανση των τραπεζών. Χρειαζόμαστε βεβαίως ένα απλό και σωστό μηχανισμό ε, για την εξυγένση των ε, τραπεζών που να μειώνει τις ε, πιθανότητες εξυγένσης ή αφαιρεγγιότητας των τραπεζών. Και οι εθνικές διατάξεις δεν θα πρέπει να αντιβαίνουν στις ευρωπαϊκές διατάξεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει αυτά τα οποία ήδη έχουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για περαιτέρω ενδυνάμωση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων MRL. Θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και θα πρέπει να μην περιορίσουμε εξ αρχής την ποιότητα των ελάχιστων απαιτήσεων μέσω των κεφαλαίων μειωμένης εξασφάλισης. Δεν θέλουμε ε, να φέρουμε κανένα πιστωτή εξ αρχής σε περισσότερο δυσμενή θέση. Όσον αφορά την αναστολή δυνατότητα πληρωμής στο μορατόριο, ε, θα πρέπει ίσως να μην ε, αποφασίσουμε εξ αρχής και η πρόταση του Γκίνερ νομίζω είναι μια πολύ καλή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Γιατί δικό μας καθήκον είναι να καταλήξουμε σε μια δέσμη μέτρων που θα καθιστά την διάσωση με ίδια μέσα ε, εφικτή και πρακτική. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ασφάλεια δικαίου, να μειώνονται οι κίνδυνοι προς όφελος ε, των ε, πολιτών που μας έχουν εκλέξει σε αυτή τη θέση. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γκούνερ και τον Πέτερ Ζήμον για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Σάντερ, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και σε πολλά σημεία συμφωνώ μαζί του. Ιδίως για το επίπεδο του ΤΙΛΑΚ και για την διάρκεια του, της ανασολής, του μαρατορίου για την εξυγένση και για την προστασία των ε, επενδυτών. Για τις απαιτήσει MRL θέλω να υπενθυμίσω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα εξυγίανσης όλων των ε, ιδρυμάτων που δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν. Θέλουμε να αποφύγουμε το να έχουμε απαιτήσει MRL και TLAC που θα επιφέρουν άνηση μεταχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με εξωτερικά πιστοτικά ιδρύματα. Και η βαθμονόμηση θα πρέπει να είναι ισορροπημένη, τηρώντας την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του επίπεδου και της ε, απαιτούμενης ποιότητας των απαιτήσεων MRL. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον εισηγητή και όλους ε, τους σκιώδεις εισηγητές που θα βοηθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε εισηγητά, φαντάζομαι ότι θέλετε το λόγο και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Χόκμαρκ. Σας ευχαριστώ όλους. Ήμουν σίγουρος ότι η αναβίωση του καπιταλισμού θα είχε μεγάλη απήχηση στην Επιτροπή μας. Ο κύριος Σόιμπλε είναι κατά του καπιταλισμού, λέει ο πρόεδρος, από ό,τι καταλάβαμε από την παρέμβαση προηγουμένως. Για διαφορετικούς λόγους ίσως. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος. Καταρχήν, για το πώς εξετάζουμε αυτή τη δέσμη μέτρων. Δεν θα έλεγα ότι είναι αναθεώρηση τη BRD. Διστάζω να πω κάτι τέτοιο για δύο λόγου. Πρώτον, διότι δεν είναι αυτό το νόημα. Δεν είναι πρόκειται για αναθεώρηση τη οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών. Δεύτερον, τώρα αγγλούμε τι εμπειρίε και τα διδάγματα από την BRD και η πραγματικότητα είναι διαφορετική σήμερα από ότι όταν αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η BRD. Διότι τότε πολλοί επενδυτές μπορούσαν να πούν ότι δεν το ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσαμε αυτόν τον κίνδυνο. Τώρα πια πολύ λίγοι θα μπορούσαν να πούν ότι δεν είχαν ενημερωθεί για τον κίνδυνο. Ήδη αυτό αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή. Και αν αυτό αποβεί πραγματικότητα θα είναι πάρα πολύ θετικό. Πολλοί συνάδελφοι λένε ότι ακόμη δεν το έχουμε καταφέρει και το καταλαβαίνω αυτό, αλλά είμαστε στη διαδικασία του να το επιτύχουμε και όσο περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι είναι περισσότερο διασώσιμα με ίδια μέσα, τόσο πιο εύκολα διασώσιμα με ίδια μέσα θα είναι. Δηλαδή όσο ε, γίνει κατανοητό και ευαισθητοποιήσουμε τους ε, επενδυτές περί αυτού, τόσο το καλύτερο. Το, άλλο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι τι θα κάνουμε με την, αναστολή, με τη δυνατότητα αναστολής πληρώματο μορατόριου. Όπως είπαμε, δεν είναι ακριβής επιστήμη αυτό το οποίο κάνουμε. Προσπαθούμε να είμαστε ρεαλιστές και να επιτύχουμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αντιτιθέμενων συμφερόντων. Θα ξαναπώ αυτό που είπα πριν, ότι θέλουμε και να είναι επιτυχημένη η εγχείρηση και να επιζήσει ο ασθενής. θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για εξυγίανση, θα πρέπει όλα τα ιδρύματα να έχουν ένα σχέδιο εξυγίανσης και αν έχουν πρόβλημα να αξιολογήσουν την κατάσταση, διότι μπορεί να υπάρχει κάποια έλλειψη στο σχέδιο εξυγίανσης και να πρέπει να εξετάσουμε μήπως τυχόν θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί έναντι των αρχών που ασχολούνται με την εξυγίανση γιατί εκείνοι θα έπρεπε να είναι πιο αυστηροί στις διατάξεις τους για τα κεφάλαια μειωμένης εξασφάλισης και το ΤΙΛΑΚ και την κατάταξη. Χωρίς να θέλω να πω ότι είναι εύκολο να κάνουμε την εξυγίανση, γιατί οι αρμόδιες αρχές δεν το θεωρούν εύκολο. Σίγουρα όμως είναι πιο εύκολο τώρα από ό,τι πριν από δύο χρόνια. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όταν συζητούσαμε το MRL ή τα υψηλότερα επίπεδα κεφαλαιακών απαιτήσεων ή τις απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης, θέλουμε κατά κύριο λόγο να εξασφαλίσουμε την οικονομική σταθερότητα. για την οικονομική σταθερότητα πρέπει να έχουμε σταθερές τράπεζες. Σε κάποια κράτη-μέλη σήμερα βλέπουμε ότι η απειλή για την οικονομική σταθερότητα δεν είναι η νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες θα σταθεροποιούσαν την οικονομία. Δηλαδή, Προσθέτοντας στις απαιτήσεις του MRL και στο TILAC και στη, σε κεφάλαια Μειωμένη εξασφάλιση κλπ. δεν βοηθάμε γιατί στο τέλος θα είναι πολύ λίγες οι επενδύσεις που θα προκύψουν από όλο αυτό το μηχανισμό. Και δική μας ευθύνη είναι να εξασφαλίσουμε την ισορροπία σε αυτό το μηχανισμό. Και ένα τέταρτο σημείο είναι ότι όπως λέμε στα σουηδικά, δεν μπορείς να τραβήξεις ε, τον εαυτό σου από τα μαλλιά. Δηλαδή, αν δεν έχουν χρήματα οι τράπεζες, κάποιος θα πρέπει να τα βρει αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε μεγάλη πειθαρχία, ώστε να τον μεγαλύτερη, να είναι όλα διασώσιμα με ίδια μέσα, διαφορετικά ξαναγυρνάμε στην αρχή. Προσβλέπω στην διεξαγωγή των συζητήσεων ε, για τη δέσμη αυτών των μέτρων και είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ επικοδομητικές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε μέσα στη δεύτερη έκθεση, στις δύο δεύτερη εκθέσεις που ακολουθούν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω γιατί με συγχαίρετε, γιατί τα έχουμε καταφέρει καλά γιατί επιβιώσαμε από τις ε, προσπάθειες. Πάντως νομίζω ότι είναι θετικό το ότι έχουμε καταφέρει σήμερα να είμαστε εδώ. Δεν έχουμε μεταφρασμένα ε, όλα αυτά τα οποία ε, έχουμε διαμορφώσει. συχνά έχουμε πολύ ε, διαφορετικές ε, καταστάσεις στα κράτη-μέλη που απαιτούν διαφορετικές λύσεις. Και υπάρχουν και εσωτερικές συζητήσεις στα κράτη-μέλη. Προσπαθήσαμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία για να λάβουμε υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και να έχουμε μια έκθεση ισορροπημένη, να λάβουμε υπόψη, βλέπω εδώ στην αίθουσα και Ιταλούς συναδέλφους και Γάλλους συναδέλφους και την ε, Σουηδική ε, κριτική όσον αφορά τις ε, κοινοτικές επιχειρήσεις και δημοτικές επιχειρήσεις. Όλα αυτά θέλαμε να τα λάβουμε υπόψη. Δέκα χρόνια μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση και τέσσερα χρόνια μετά την ε, ε, ενιαία δέσμη μέτρων για τη ρύθμιση των τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προτείνει τώρα κάτι καινούριο. Βλέποντα λοιπόν αυτό που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπουμε ότι θέλουμε και την ε, μείωση των κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και χρηματοδότηση της οικονομίας και αναλογικότητα και ρύθμιση των τραπεζών. Ας ξεκινήσουμε με τον κίνδυνο ε, και με το δίκτυ μόχλευσης. 3% προτείνει η Επιτροπή, το θεωρώ σωστό, αλλά για τα g γιατί έχουμε, να έχουμε 3% δίκτυ μόχλευσης. Στην πράξη όλες οι μεγάλες τράπεζες ε, ήδη σήμερα ε, το έχουν επιτύχει αυτό και διαπιστώνουμε ότι σε άλλες χώρες όταν θέλουμε να έχουμε ε, συνθήκες ίσου ανταγωνισμού και δίκαιου ανταγωνισμού, βλέπουμε ότι σε πολλές χώρες έχουμε υψηλότερο δίκτυ μόχλευσης. Παραδείγματος χάριν, στις ΗΠΑ ή στην Ελβετία, βλέπουμε 5%, 6%. Θα μου πει κάποιος ότι οι κίνδυνοι ε, για τα ενυπόθηκα ε, δάνεια της φανή μέη βγήκαν από τα βιβλία. Αυτό και ισχύει και δεν ισχύει. Διότι ναι μεν ισχύει, αλλά αν τα προσθέσετε αυτά, στις ΕΠΑ φτάνουμε σε δίκτυ μόχλευσης 4%. Γιατί ο κίνδυνος της Fannie Mae, της Freddie Mac ήταν γύρω στο 1%. και νομίζω ότι υπάρχει διεθνής υποστήριξη για μια αύξηση του δίκτυ Για τις άλλες ε, ε, συστημικά σημαντικές τράπεζες προτείνεται μια προσαρμογή που δεν θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που ζητείται από τις παγκόσμιες συστημικές ε, τράπεζες. και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι κυκλικοί κίνδυνοι. Τα αντικυκλικά αποθέματα είναι απαραίτητα για να μπορούν να αντίσταται οι τράπεζες ε, στους κινδύνους ε, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη χορήγηση πιστώσεων στην πραγματική οικονομία. τράπεζες που έχουν ε, πιο αυστηρές απαιτήσεις δεν θα χρειάζεται να δημιουργήσουν επιπλέον κεφάλαιο. Αυτό το οποίο προτείνεται εδώ ως προσαρμογή στην έκθεση είναι ότι θα πρέπει να έχουμε προσαυξήσεις κεφαλαίου όταν αυξάνεται το αντικυκλικό απόθεμα. Στην ε, έκθεσή της η Επιτροπή μιλά και για το δίκτυ καθαρής σταθερής χρηματοδότησης. εάν ε, αυτό μπορεί να γίνει βραχυπρόθεσμα, αλλά πιο μακροπρόθεσμα, Χρειαζόμαστε το δίκτυο καθαρή σταθερή χρηματοδότηση Για μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση, ούτως ώστε να υπάρχει επαρκής ρευστότητα για ένα χρόνο. Στην έκθεσή μου προτείνω κάποιες συγκεκριμένες ε, αλλαγές στο δίκτυο καθαρής σταθερής χρηματοδότησης χωρίς να αλλάζουμε τη γενική έννοια. για την ε, αναχρηματοδότηση παραγόγων, παραδείγματος χάρη, προτείνουμε μια μείωση από το 20% στο 15% και για τα υπόλοιπα παράγωγα να το αφήσουμε στο 10%. Τις απαιτήσει ε, εξισορρόπησης τις αφήνουμε απαράλλεκτες. Προτείνεται μια απλουστευμένη, ένας απλουστευμένος δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότης NSFR για τις μικρότερες ε, ε, τράπεζες. Μια ε, απλουστευμένη εκδοχή του NSFR με 10% όταν υπάρχει και αυστηρότερη βαθμονόμηση για να έχουμε παρόμοιες ε, απαιτήσεις εποπτικής εξέτασης. Διευκολύνονται λοιπόν οι μικρότερες τράπεζες χωρίς να φύγεται η προληπτική εποπτεία. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει επίσης και το θέμα της αναθεώρησης του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους σε μεγαλύτερο βαθμό μια αρχική περίοδος δύο ετών και μετά άλλα τρία χρόνια με 65%. Στην έκθεσή μου το προσαρμόζω αυτό για να μην έχουμε κάποιες αδυναμίες που θεωρούμε ότι έχει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιμηκύνω τη φάση υλοποίησης από τα δύο στα τρία χρόνια για να μπορέσουμε ε, να διαμορφώσουμε τις απαιτούμενες τεχνικές ε, διατάξεις και αυτό δίνει και μεγαλύτερη ευελιξία στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προετοιμαστούν. Δεν έχω πλέον χρόνο. Δούλεψα τόσο πολύ και δεν έχω χρόνο να τα παρουσιάσω. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχω να πω. Θα μπορούσα και να σταματήσω εδώ, αλλά ε, την, ε, να, θα, σας τα πω μονολεκτικά. Νομίζω ότι είχα ένα τέταρτο, αλλά δεν έχω. Ε, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, τα τρία χρόνια θα περνούσαμε ε, από το 65% στο 100%. Στα πέντε χρόνια που προβλέπω εγώ, αρχίζουμε από το 60% και προσθέτουμε 10% το χρόνο. Οπότε έχουμε μια σταδιακή προσαρμογή για να μην υπάρχει το cliff effect που υπάρχει στην ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, όσον αφορά ε, τις ε, αποδοχές, κάτι παρόμοιο με την Αμερικανική νομοθεσία. Δηλαδή, εισάγουμε ένα ποσοστό το οποίο ορίζει μόνη της η κάθε τράπεζα. Αποφασίζει τα θέματα αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας κάποιο ποσοστό της αμοιβή των υπαλλήλων. Αλλά θα πρέπει αυτό το ποσοστό το οποίο ορίζει ως αποδοχές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να το δημοσιοποιεί. Κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για τις αμοιβέ των ε, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με, τις, ε, ε, με τα συμπεράσματα της ομάδας δράσης για το κλίμα, λαμβάνουμε υπόψη και θέματα βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινδύνων. Δηλαδή όταν μια τράπεζα αναλαμβάνει δεσμεύσεις για τη βελτίωση του κλίματος, θα πρέπει και αυτό να λαμβάνεται υπόψη και να λαμβάνονται υπόψη και οι κίνδυνοι για το κλίμα. Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα τα οποία θα μπορούσαμε να δώσουμε. Επενδύσεις σε υποδομές μιλάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της ε, για αναχρηματοδότηση επενδύσεων, έργα υποδομών τα οποία διεξάγονται από ιδιωτικές εταιρείες για τις οποίες παρέχονται εγγυήσεις από δημόσιους οργανισμούς. Δεν νομίζω ότι συμφωνούμε με την προσέγγιση αυτή και εδώ θέλουμε να εξασφαλίσουμε ίση μεταχείριση. Μιλάμε για επενδύσεις σε υποδομές, ακόμη και αν αυτές οι υποδομές διεξάγονται από δημόσιους φορείς. και δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν έσοδα, δηλαδή στους αυτοκινητοδρόμους μπορεί να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν διόδια. Όταν θέλουμε τις υποδομές να τις κρατήσουμε χαμηλού κόστους. Και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πιστώσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προτείνουμε ένα πράσινο παρονομαστή, δηλαδή διευκολύνονται οι επενδύσεις σε πράσινα περιουσιακά στοιχεία ή σε έργα φιλικά προς το κλίμα. Τέλος, για την ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων. Ε, και εδώ διευκολύνονται οι επενδύσεις όταν ο ε, επενδυτής προσφέρει κάποιες εγγύσεις, οπότε μειώνεται ο κίνδυνος των τραπεζών. Κλείνοντας για την αναλογικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διευκολύνουμε την κατάσταση για τις μικρότερες ε, ε, τράπεζες. με την πρότασή της η Επιτροπή πιστεύω ότι δεν προσπαθεί, δεν φτάνει όσο θα θέλαμε ε, να προχωρήσει. Ε, υπάρχουν και κάποια ποσοστά ε, της, ε, του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ίσες συνθήκες ε, στη Μάλτα και στη Γερμανία παραδείγματος χάρη όπου το ΑΕΠ είναι εντελώς διαφορετικό. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τον ορισμό των μικρών και μη πολύπλοκων ιδρυμάτων και όταν μιλάμε για 1,5 δις ισολογισμού, να προσθέσουμε ένα συντελεστή 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αλλά δεν αντικατοπτρίζεται το προφίλ κινδύνου για τα μικρά και μη πολύπλοκα ιδρύματα. Θέλει η Επιτροπή να δώσει κάποιες ελαφρύνσεις προς ε, τα μικρά ιδρύματα. ελαφρύνσεις ε, για το διοικητικό κόστος μπορεί να δίνονται και μέσω μιας ε, απλοποιημένης αλλά πιο αυστηρής βαθμονόμησης του NSFR, του Δίκτυου Καθαρής Σταθερής ε, Χρηματοδότησης και θα μπορούσα να σας πω πολύ περισσότερα για την αναλογικότητα αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει περισσότερη υπομονή ο Πρόεδρος οπότε περιορίζομαι σε αυτά και θα πούμε πολύ περισσότερα στις μελλοντικές μας συνεδριάσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικά δύσκολο ήταν για σας να συνοψίσετε σε τόσο λίγα λεπτά μια τόσο εμπεριστατωμένη έκθεση και μακροσκελή, αλλά πρέπει να κλείσουμε στις 9.30 και και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να πάρουν το λόγο όλοι οι σκιώδεις εισηγητές. Ξεκινάμε με τον κύριο Κάρα, εισηγητή από πλευράς ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή που μας έκανε την παρουσίαση της έκθεσης. Σε τρία σημεία θέλω να κάνω κάποια σχόλια. Για τον τομέα της αναλογικότητας, μόνο σε κάποιες λεπτομέρειες χρειάζονται κάποιες τροποποιήσεις. Μέχρι τις 25 Ιανουαρίου έχουμε χρόνο για την υποβολή τροπολογιών. Και θα γίνουν πολλές συζητήσεις με τους συναδέλφους. Καλό θα ήταν να γίνουν συζητήσεις για να ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση κινούμεθα. Ε, συμφωνώ με τον ορισμό για τα μικρά και μη πολύπλοκα ιδρύματα όπου μπορεί να δοθούν ελαφρύνσεις. Ε, επίσης, ε, τα θέματα της αναλογικότητας για τον κίνδυνο αντισυμβαλωμένου με βρίσκουν σύμφωνο. και για τη μείωση του κόστου συμμόρφωσης των μικρών και μη πολύπλοκων ιδρυμάτων επίσης είμαι σύμφωνος. Θα πρέπει να βρούμε συνέργειες με το πλαίσιο του 2015 ε, όσον αφορά και ε, τις ε, αποδοχές θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις εθνικές διατάξεις για να μην έχουμε ένα κατακαιρματισμό των μέτρων τα οποία προτείνονται. Στα πλαίσια του πυλώνα 2 υπάρχουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι για συγκεκριμένα πιστοτικά ιδρύματα και πρέπει να βρεθεί σωστή ισορροπία μεταξύ της ευελιξίας ε, ε, ε, για εθνικές ιδιαιτερότητες και του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τα συνολικά πρότυπα και τη μείωση κινδύνου Πιστεύω ότι για το δίκτυ μόχλευσης ε, για τα συστημικά ιδρύματα είναι δικαιολογημένο αυτό το οποίο προτείνεται και στην Βασιλεία προτείνεται για την ε, βαθμονόμηση και την υλοποίηση που σύμφωνα με τη Βασιλεία το 2020 θα υλοποιηθεί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις συνολικές προτάσεις και είναι δικαιολογημένες οι προσαρμογές του δίκτυ μόχλευσης. Όσον αφορά το δίκτυ καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, επίσης κινούμεθα προς την ε, σωστή κατεύθυνση. Για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών πρέπει να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ευρώπη τηρεί τις υποχρεώσεις της και χρειαζόμαστε μια αναλογική ε, προσαρμογή ε, όπως ε, πρότεινε ο εισηγητής. ώστε να μην έχουμε υπερβολική νομοθέτηση. Ούτε θέλουμε να έχουμε υπερβολικές διατάξεις και υπερβολικές αντιδράσεις. Κάτι το οποίο πάντοτε ε, μου είναι προσφυλές ε, είναι το θέμα των πράσινων περιουσιακών στοιχείων και της υποστήριξης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Σε αυτή την έκθεση δεν καταλαβαίνω όμως πώς ταιριάζει αυτή η έννοια. Έχουμε κάποια βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των ε, κινδύνων και δεν βλέπω να υπάρχουν στοιχεία ότι για, τις, ε, ε, για τα πράσινα περιουσιακά στοιχεία είναι περιορισμένος ο κίνδυνος. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο συγκεκριμένα τεκμήρια και για τις ε, κοινωνικές επιχειρήσεις. Αν έχουμε κάτι το οποίο είναι μετρήσιμο, θα συμφωνήσω. Αλλά αν είναι κάτι το οποίο δεν είναι μετρήσιμο, ε, ε, πώς θα το βάλουμε κατευθείαν σε μια κατηγορία χαμηλότερου κινδύνου. Ίσως ε, χρειάζεται λίγο περισσότερη επεξεργασία αυτό το θέμα. Επίσης, ένα άλλο θέμα για τη δημοσιοποίηση ε, του ποσοστού αποδοχών οι αποδοχές ε, δεν θα πρέπει να δημιουργούν ένα επιπλέον κριτήριο κινδύνου. Θέλουμε να έχουμε διαφάνεια και να λαμβάνονται υπόψη και τα μπόνους τα οποία δίδονται από τις τράπεζες. Άλλα θέματα τα οποία ίσως πρέπει να αναφερθούν είναι θέματα επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες όταν η μητρική εταιρεία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ψηφιοποίηση συνεχίζεται, χρειάζεται να έχουμε σαφήνεια. Και όσον αφορά την έκθεση, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν. και να υπάρχει ώστε να τον μεγαλύτερη σαφήνεια. Κάποια σημεία δεν αναφέρονται, ενώ στη Βασιλεία αναφέρονται και θα μπορούσαν και εδώ να συμπεριληφθούν. Ευχαριστώ τον εισηγητή και θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε μέχρι ε, την προθεσμία υποβολής τροπολογιών και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τις καλύτερες δυνατές συμβιβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φόξου για το ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθώ να παραμείνω σύντομος, όπως με ακολουθεί η φήμη μου άλλωστε. Ευχαριστώ τον κύριο Σάιμον για την έκθεση. Η ομάδα μου πιστεύει ότι είναι βελτίωση σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Πρέπει να ανταγνωρίσουμε τη Συμφωνία της Βασιλείας τη περασμένη εβδομάδα και να εργαστούμε σε αυτό το πλαίσιο. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει να εφαρμόσει τους κανόνες για του κινδύνου τη αγορά μέχρι το 2022 και να έχει τους απαραίτητους κανόνες για να συνεχίσει την απαραίτητη τεχνική εργασία. Για το δίκτυο με μόχλευση οι του εισηγητή είναι πολύ σημαντικέ, αλλά και για το δίκτυο καθαρή σταθερή χρηματοδότηση, ένας παράγοντα του 5% θα είναι βοηθητικό από τη στιγμή που του χρόνου θα ολοκληρωθεί και η δουλειά για τα παράγωγα. Από εκεί και πέρα. Θα ήθελα να μιλήσω για το πλαίσιο της αναλογικότητας. Ο εισηγητή δείχνει δεσμευμένο στην αρχή της αναλογικότητας σε όλο το κείμενο και αυτό είναι ευπρόσδεκτο. Βεβαίως αυτό βοηθά την ειδική γερμανική τραπεζική δομή και θα πρέπει να επεκταθεί κι αλλού. Πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να φανεί και στα κατόφλια για την εφαρμογή στο άρθρο 90 της πρότασης της Κομισιόν. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να θέτουν τα κατόφλια, κατόφλια και αν τα ξεπεράσουν οι, οι τράπεζες θα πρέπει να υπόκεινται στους κανόνες τους εγχώριους για την αμοιβή εννοώ και τις αποδοχές. Από εκεί και πέρα, το Intermediate Parent Undertaking. Ε, με εκπλήσι που η Κομισιόν προτείνει IPU χωρίς αξιολόγηση αντικτύπου και έχουν γίνει αλλαγέ. Αυτό είναι πολύ λυπηρό. Πώ θα αξιολογήσουμε το κατά πόσο δρούμε αναλογικά, ενώ δεν έχουμε λεπτομερή ανάλυση. Ε, στοχεύουμε τι σωστέ τράπεζε, πιάνουμε τι σωστέ τράπεζε και τι θα γίνει με τα διεθνή GSIB που δεν έχουν στοιχεία ενεργητικού 30 δις ευρώ εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά θα του διώξουμε του επενδυτέ αυτού και θα χάσουμε τις θέσεις απασχόληση που θα δημιουργούσαν. Να δούμε το διεθνέ πλαίσιο. Δεν μιλούμε μόνο για τι αμερικάνικέ τράπεζες. Δεν εγκρίνουμε τις διασυνοριακές ε, ε, προληπτικές εξαιρέσεις waiver γιατί αποκλίνουν από τους κανόνες CRTV αλλά και δεν ωφελούν και σε τίποτα από τους κανόνες του κανονισμού δηλαδή για τις απαιτήσει για ίδια κεφάλαια. Και θα θέλαμε τη διαγραφή αυτής της αναφοράς. Τώρα για τους παράγοντες έκπτωσης, discount factors, ίσως έχει κάποια αξία αυτό, αλλά πρέπει να δουλέψουμε περιττέρω, να διασφαλίσουμε ότι όντως λειτουργεί. Ε, και ο ορισμός της πράσινης χρηματοδότησης είναι δίσκαμπτος αυτή τη στιγμή. Το μήνυμα μας, κύριε Σάμιον είναι το εξής. Βελτιώσατε αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εμείς θέλουμε να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η Καρολίνα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και εγώ με τη σειρά μου για τη δουλειά του ε, και ελπίζω ότι θα βάλουμε όλοι ένα λιθαράκι για την υιοθέτηση της θέσης του Κοινοβουλίου. Και ε, χαίρομαι και για την καθυστέρηση στην εξέταση όλων αυτών, γιατί μπόρεσα αυτέ τι εβδομάδε να εγκατασταθώ και να καταλάβω περίπου τι γίνεται. Νομίζω ότι τι διακοπέ των Χριστουγέννων θα τι περάσω ασχολούμενοι με αυτά τα θέματα επισταμμένω. Τι πρώτε μου εντυπώσει όμως θα σα τι πω σήμερα. Το τραπεζικό ε, πακέτο είναι η δέσμη μέτρων η πιο σημαντική σε ό,τι αφορά τα θέματα συναπόφασης. Ε, και η μείωση του κινδύνου είναι ακρογωνιαίος λήθος για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και ο κανονισμός για τις απαιτήσει σε ίδια κεφάλαια, η οδηγία, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Οι κατευθυντηρίες γραμμές όπως αυτές της Βασιλείας αποτελούν τη βάση μεγάλου μέρους της νομοθεσίας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η διεθνή συνεργασία είναι απαραίτητη για να έχουμε ένα αθεκτικό και σταθερό χρηματοπιστωτικό τομέα. Η Επιτροπή της Βασιλείας και άλλα όργανα συμβάλλουν σημαντικά, σημαντικότατα και ελπίζω και θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν θα αλλάξει. Την περασμένη εβδομάδα κατέστησε σαφές ότι οι προτάσεις της Βασιλείας δεν είναι όλες ισορροπημένε. Δεν... Το ελπίζαμε, αλλά δεν συνέβη. Βεβαίως η διεθνή συνεργασία είναι απαραίτητη. Ένα παιχνίδι επίσης όρου μεταξύ Ευρώπη και άλλων χωρών θα πρέπει να είναι και η βάση για αυτή τη συνεργασία. Άλλωστε, τα επόμενα χρόνια θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτού του είδους τη συνεργασία αναμένοντας και την επόμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα δεν σας εκπλήξει, δεν θα σας εκπλήσει το γεγονός ότι εγώ δεν είμαι υπέρ υψηλότερων κεφαλαϊκών απαιτήσεων για τις μεγαλύτερες τράπεζες. Για να είμαι ειλικρινής, όμως άκουσα τις εξηγήσεις σας προλίγου, προσπαθήσατε να με πείσετε μην πανηγυρίσετε γιατί δεν το καταφέρατε 100% αλλά εν πάση περιπτώσει ανοίγει ένα περάθυρο για να το συζητήσουμε λίγο μεταξύ μας περισσότερο. Πράγματι είναι σημαντικό να είναι ανθεκτικός ο χρηματοπιστωτικός τομέας αλλά είναι σημαντικό και να έχουμε ένα παιχνίδι επί ίσης όρης. Να είμαστε προσεκτικοί όταν θα βρούμε το σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ των δύο. Και ελπίζω και προτιμώ αυτό να γίνει σε διεθνές επίπεδο και όχι εντό Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η προσυζήτηση είναι αυτό. Σημειώνω τι τροπολογίε του κυρίου Σάιμον για την αναλογικότητα και είναι μια αρχή που μα βρίσκει σύμφωνο. Πρέπει να προσπαθήσουμε όμω και εδώ να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπίας και να μην δημιουργήσουμε νέα σημεία ευαλωτότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Για μένα ως Ολλανδή ε, η αντιμετώπιση των mortgages είναι πάρα πολύ σημαντική, υποθήκες κλπ. Καλωσορίζω την τροπολογία 61 του εισηγητή, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, παρόλο που μπορεί να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω και έτσι το μοίρασμα του κινδύνου να γίνει πιο σωστό και πιο δίκαιο. Τώρα, οι διατάξεις για τις αποδοχές ίσως αποδειχθούν πάρα πολύ ευαίσθητες, δηλαδή να περιοδοτήσουν ζητημάτα πολύ λεπτά και ιδίω ε, σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινή γνώμη. Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν νέα στοιχεία που μπαίνουν στο παιχνίδι, κοινωνικοί παράγοντες, ε, πράσινη ανάπτυξη, κλιματικά θέματα και πρέπει να τα συζητήσουμε. Εγώ και η ομάδα μου θα εργαστούμε πάνω σε αυτά, αλλά και για το θέμα του software και του free flow με τις promotional banks. Περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να συνεργαστούμε για να συμβάλλουμε σε έναν αθεκτικό και ανταγωνιστικό όμως χρηματοπιστωτικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η συζήτηση στην Επιτροπή μας. Ο Ματ Κάρθ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο εκθεσής του. Ε, καλωσορίζουμε τις ιδέες που έχει παρουσιάσει και πιστεύουμε ότι μικρότερες και, λιγό... και τράπεζες που έχουν λιγότερους κινδύνους θα πρέπει να τύχουν διαφορετική μεταχείριση σε σύγκριση με τις συστημικώς σημαντικές. Εμείς έχουμε ανέκαθεν ταχθεί υπέρ των μικρών τραπεζών που να μπορούν να εξηγηθούν αρκετά εύκολα χωρίς να συμβάλλουν οι φορολογούμενοι Άρα, η δέσμη αυτή μέτρων ε, πρέπει να μπορέσει να συμβάλλει σε ένα σωστό και ισορροπημένο τραπεζικό σύστημα και θα πρέπει να μειωθεί ο κίνδυνος του τραπεζικού τομέα. Οι μεγάλες τράπεζες να γίνουν μεγαλύτερες, να γίνουν μικρότερες, συγγνώμη. Και καλωσορίζουμε τις προτάσεις της Κομισιόν που αποκλίνουν από τα πρότυπα της Βασιλείας εφόσον συμβάλλουν να ε, ε, αναζωογονήσουν και να ενθαρρύνουν την πραγματική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ισχύει. Πολύ το αμφισβητώ. Πιστεύουμε ότι η δέσμη αυτή μέτρων πρέπει να εστιάζει την προσοχή της στις συστημικό σημαντικές τράπεζες και παγκοσμίως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το too big to fail, οι τράπεζες που είναι υπερβολικά μεγάλες για να καταρρεύσουν πρέπει να λυθεί επιτέλους. Και γι' αυτό ελπίζουμε να συνεργαστούμε με τους κυριώδες εισηγητές για να τροποποιήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δίκτυο μόχλευσης. Συμφωνούμε με τον εισηγητή. Είναι πολύ χαμηλό για τις παγκοσμιοσυστημικές ε, σημαντικές ε, τράπεζες. Και θέλουμε ο συντελιστής να είναι τουλάχιστον 5% και θα ε, θα έχει διπλάσια ωφέλη σε σχέση με το 3%. Η Επιτροπή θέλει να απαλλάξει κάποια στοιχεία από το δίκτυο μόχλευσης. Εμείς δεν συμφώναμε με αυτές τις παρακλήσεις ή εξαιρέσεις και θα πρέπει να υπάρχουν συστάσεις για τη βαθμονόμηση του δίκτυου μόχλευσης. Η αύξηση 4% που προτείνει ο δεν είναι αρκετά υψηλή. και θα δούμε και τις προτάσεις για τις promotional banks και τις προωθητικές τράπεζες και τις προωθητικές ε, δράσεις γενικότερα. Σε κάθε περίπτωση το υφιστάμενο TILAC, η συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών, δεν είναι αρκετή για να απορροφήσει τους κραδεσμούς από την επόμενη τραπεζική και ε, χρηματοπιστωτική κρίση μόνο οι, οι, πιο, οι τράπεζες που είναι πιο ψηλά στην ιεραρχία, στην, στο πλαίσιο της βασιλείας, θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο ΤΙΛΑΚ. Επομένως, ότι θα τεθούν πολλά ερωτηματικά για τις υπόλοιπες και κατά πόσο θα μπορέσουν να εξηγιανθούν με ασφάλεια. Οι αποτεχίες των συστημικών σημαντικών τραπεζών θα έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα. Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 19,2 για να περιλαμβάνει ε, ελάχιστες απαιτήσει σε ίδια κεφάλαια και για τις OS2 ε, και GS3, δηλαδή τις σημαντικές για το σύστημα, τα σημαντικά για το σύστημα ιδρύματα αλλά και τα σημαντικά για το παγκόσμιο σύστημα ε, τραπεζικά ιδρύματα. Η εξαίρεση για το σημείο 11 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί υπάρχει κίνδυνος ε, που έχει να κάνει με τις νομικές προκλήσεις. Τώρα στο άρθρο 501β Νομίζω ότι το περιεχόμενό του δεν ταιριάζει σε όλες τις τράπεζες. Πρέπει να έχουμε ένα scaling factor και να έχουμε 40% για τους μεν και 80% για τους δε. Και να έχουμε μια περίοδο σταδιακής εισαγωγής όλων αυτών εντός τριών ετών θα υποβάλουμε τροποποιήσεις στις τροπολογίες 64 54 με 65, αλλά και θα ζητήσουμε διευκρινήσεις και για το δεύτερο πυλώνα και τις ε, κατευθυντηρίες γραμμές για τα κεφάλαια δεν θα πρέπει να εξασθενήσουν οι αρμοδιότητες εποπτείας και δεν θα πρέπει να περικοπεί το περιθώριο έλιγμων ε, και χειρισμών της ελεγκτικής αρχής και της αρχής εποπτείας. Είμαστε κατά της διαγραφής του άρθρου 103 του CRD4 όπου μιλάμε για το μακροπροληπτικό πλαίσιο. Και για το άρθρο 341 δεν βλέπουμε λόγο να υπάρχουν οι εξαιρέσεις στο δεύτερο εδάφιο. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε βάθος με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Σβεν Γκίγκολ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω γερμανικά και θα συνεχίσω αγγλικά. Στα γερμανικά θα σας πω ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ στον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης που σε γενικές γραμμές την υποστηρίζουμε. Σας ευχαριστώ διότι προσπαθήσατε να υποστηρίξετε και τις δικές μου προτάσεις Όσον αφορά τις ημερομηνίε ε, και την ε, λάβατε υπόψη τι ε, προτάσεις μου. Πέρα τούτου, αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι μετά από 10 χρόνια, μετά από 10 χρόνια κρίσης, τι κάναμε σωστά και τι λάθος. Ξέρω ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης της επίσημης, διάφορες ομάδες και διάφοροι βουλευτές ε, αρέσκονται σε κάποια τμήματα του καπιταλισμού. Είναι ε, ενδιαφέρον να βλέπει κανείς ότι η αντίληψη του καπιταλισμού μπορεί να βελτιωθεί και στην αριστερά. Έχουμε το ΕΛΚ επίσης, το οποίο δίνει μάχη για κάποιες άλλες πτυχές του καπιταλισμού και η σοσιαλιστική οικογένεια επίσης έχει αυτή μια ιδιαίτερη στάση ενώπιον του καταπερισμού ανάγω με τη χώρα μέλος και τον βουλευτή. Και το παράξενο και με εμά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τεράστιες εθνικές διαφορές. Στην έκθεση πάντως, εκεί που συμφωνούμε απολύτως, είναι ότι χρειαζόμαστε παντού αναλογικότητα. Και αυτό νομίζω είναι και η βασική ιδέα που ακολουθεί ο συγητής. Όσον αφορά την αναλογικότητα προς τα κάτω, θα πρέπει να πω ότι εμείς υπερθεματίσαμε κάποιους φορείς με υποχρεώσεις υποβολής έκθεσης. Δεν είναι γερμανικό θέμα ή βρετανικό θέμα. Όλοι παραπονιούνται γι' αυτό, ότι δηλαδή δημιουργήσαμε κανόνες οι οποίοι είναι υπερβολικοί και που δεν έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην χρηματοοικονομική σταθερότητα. Οπότε η βασική γραμμή του εισηγητή είναι ότι εμείς ακριβώς δεν θα αντιμετωπίσουμε θέματα χρηματοοικονομικής σταθερότητας μέσω δικτών ή μέσω αυτού που είπε και ο κύριος Καράς, αλλά αντίθετα θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στο βάρος και με αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Θεωρώ λοιπόν ότι σε κάποια ζητήματα μπορούμε να προχωρήσουμε και είπαν διάφοροι κατηδίαν ότι το πρόβλημα δεν είναι το απόλυτο βάρος αλλά η ταχύτητα των αλλαγών που έχουν θεσπιστεί. Γιατί λοιπόν τουλάχιστον αν δεν υπάρχει επίγον ή κατεπίγον να μην πούμε ότι σε ένα-δύο χρόνια να θεσπίσουμε νέα υποχρέωση υποβολής έκθεσης ώστε να προσαρμοστούν, να μπορούν να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος one-stop shop όσον αφορά την υποβολή των εκθέσεων. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που είπε και ο κύριος Κάρας. Δηλαδή η υποπτική αρχή και η στατιστική αρχή θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται και να συγκλίνουν όσον αφορά την υποβολή των εκθέσεων από τους μικρότερους, ώστε το βάρος δηλαδή της υποβολής να είναι πιο μικρό. Πέραν τούτου, είμαστε πεπισμένοι ότι οι μικρές τράπεζες, οι οποίες δεν θα πάνε σε εκαθάριση, αυτές θα επιβαρηθούν από πολύ λεπτομερή σχέδια εξεγένσης. Θεωρούμε ότι θα μπορούσε να αρκέσει αντί να έχουμε πολύ περίπλοκα έμρελ να τις απαλλάξουμε τις τραπέζες αυτές από αυτά αν η αντίστοιχη, το αντίστοιχο ίδρυμα ήδη διαθέτει κάποια κεφάλαια. Και τέλος, δεν καταλαβαίνουμε γιατί οι μικρές και υγιείς τραπέζες χρειάζονται κίνητρα για τα παράγωγα, όπως ακριβώς αναφέρουν οι υδροπολογίες 75 και 76. Θέλουμε εδώ περιττέρω εξηγήσει. Πέραν αυτών, όσον αφορά τώρα την αναλογικότητα προς τα πάνω, συμφωνούμε με τον εισηγητή όσον αφορά την αύξηση του δίκτυ μόχλευσης για τα G-SIPS. Συμφωνούμε επίσης ότι θα πρέπει να έχουμε δεσμευτική και πιο βαθμιαία αναθεώρηση του βιβλίου συναλλαγών και να συζητήσουμε εδώ βέβαια τις ε, λεπτομέρειες αλλά για τη γενική κατεύθυνση συμφωνούμε. Επίσης να πω ότι δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι σημαντικό σχετικά με αυτό και έχουμε και σοβαρές αφιβολίες σε σχέση με ε, τις εμπορικές τράπεζες ώστε να μην έχουμε τριβές σε σχέση με αυτές τις τραπέζες. Και θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν αποκλίνουμε από τα πρότυπα της Βασιλείας όσον αφορά το τίλακ. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι όταν εφαρμόζουμε εθνή πρώτα ότι γινόμαστε πιο δυνατοί. Επίσης της τραπεζές. Εδώ θα έχουμε, πρέπει να έχουμε κάποιους περιορισμούς και τουλάχιστον να περιοριζόμαστε στο καθεστώς ανοιγμάτων ώστε ακριβώς να καταπολεμήσουμε τις επικίνδυνες διασυνδέσεις τραπεζών και κυβερνήσεων. Επίσης θα ήθελα να πω και δύο λόγια σχετικά με τους διάφορους ε, υποστηρικτικούς παράγοντες. Συμφωνούμε απολύτως για το ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αξιολογούν κλιματικούς παράγοντες και άλλους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό να γίνεται συστηματικά από όλες τις τράπεζες, ώστε με τη σειρά της η αγορά, και εδώ κάπως διαφέρω από αυτό που ο Ότμαρ Κάρας προηγουμένως, ώστε οι αγοράς ακριβώς να μπορέσουν να κεφαλοποιήσουν αυτούς του κινδύνους και να υπάρχει διαφάνεια. Από την άλλη μεριά, έχουμε αφιβολίες σε σχέση με όλα αυτά τα υποστηρικτικά στοιχεία και παράγοντες. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Μας λένε ότι υπάρχουν κεφάλαια. Υπάρχουν κεφάλαια, αλλά κίνδυνοι δεν αποτιμούνται επαρκώς. Και ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολύ λίγα προγράμματα, λίγα projects, ε, ΑΠΕ ας πούμε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που δεν ε, χρηματοδοτούνται αν δεν έχουν τις κατάλληλες, ε, τα κατάλληλα κέρδη. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογισμό κινδύνου χωρίς πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία ότι κάτι είναι λιγότερο επικίνδυνο, παρουσιάζει λιγότερους κινδύνους. Θα πρέπει να δούμε ας πούμε αν αυτό έχει να κάνει με την κοινωνική οικονομία ή με, την, με το λιανικό εμπόριο στεγαστικών δανείων. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τον υπολογισμό κινδύνου και το κεφαλαϊκό βάρος. Παρόλο που μπορεί να υπάρχουν καλές προθέσεις, μπορούμε τελικά να χάσουμε αυτούς τους ε, παράγοντες που έχουμε στον, ε, στην νομοθεσία για σωστούς λόγους. Αν θέλουμε, λοιπόν, αν θέλουμε και επιθυμούμε περισσότερη πράσινη χρηματοδότηση, να δούμε τι γίνεται με τις απαιτήσει που ήδη έχουμε και τα εργαλεία που ήδη διαθέτουμε και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να κάνουμε από τώρα. Δεν είναι πρόημο και είμαστε υπέρ απολύτως του να γίνει κάτι τέτοιο. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πω ότι έχει κάνει επανειλημμένω μια έκκληση. Ναι, τελειώνω πρόεδρε. Να σταματήσουμε με αυτές τις εθνικές επιλογές και διακριτικές ευχέρειες. Ο εισηγητής είπε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα σοβαρά την σύσταση αυτή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπέζα και να κάνουμε τις αλλαγέ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, για τα στεγαστικά, αυτό το θέμα βρίσκεται στο πακέτο τη Βασιλεία. Έτσι και συμφωνώ εξάλλου απόλυτα μαζί σα, λέει ο πρόεδρο. Ο Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και εγώ συγχαίρω τον Πίτερ Σίμον, τον εισηγητή, για τη δουλειά που έκανα. Και πρέπει να πω ότι η δουλειά ήταν καλή Παρόλο που δεν συμμεριζόμαστε τα πάντα, θεωρώ ότι όντως θα πρέπει να αποφεληθούμε το Χριστουγέννο γιατί είμαστε μόνο στο 10% αυτών πρέπει να γίνουν. Να πω δύο λόγια σύντομα γιατί έχουμε ένα κανόνα ενιαίο ο οποίος θα πρέπει να εφαρμοστεί σε τράπεζες χωρίς να έχουμε πραγματική Τραπεζική Ένωση και ήδη αυτοί οι κανόνε μέχρι τώρα έχουν δημιουργήσει μεγάλη συμμετρία μεταξύ των διαφορών τραπεζικών συστημάτων στην Ευρώπη. Οπότε το να εφαρμόσουμε νέου κανόνε ξαφνικά χωρί να λάβουμε υπόψη μα τι επιπτώσει, θα οδηγήσει κάτι τέτοιο σε πολλέ ανισορροπίε σε χώρε οι οποίε ήδη έχουν πληγεί από την κρίση και έχουν πολύ ευαλωτή ανάπτυξη Όπω η δική μου χώρα η Ιταλία που έχει μια ένα, ένα τραπεζικό σύστημα που στηρίζεται στην πίστοση. Οπότε χαίρομαι που ο εισηγητής θέλει να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις όπως και την ανισορροπία που έχει παρεσφρήσει σε θέματα όπως η πίστοση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υποπτέψουμε τον κίνδυνο το χρηματοοικονομικό όσον αφορά την κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών. Θέμα πολύ σημαντικό γιατί την επόμενη συστημική κρίση θα την ε, πληρώσουμε όλοι και ιδιαίτερα μέσω ρευστών, μέσω ρευστού γιατί ακριβώς έχουμε επικεντρωθεί στην πίστοση. Για την έκθεση λοιπόν συμφορούμε με το δίκτυο μόχλευσης η Κομισιόν προτείνει 3%, ο εισηγητές 4%, εμείς θέλουμε περισσότερο ακόμα 5% ως δεκτημόχλευσης, αλλά νομίζω θα βρούμε μια λύση. Συμφωνούμε επίσης και με τις ε, παρεκκλήσεις όσον αφορά τις απαιτήσει. Αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην πιέσουμε την πίστοση. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια αγορά κεφαλαίων που δημιουργεί πολλές ευκαιρίες αλλά ταυτόχρονα και πολλές καταστάσεις όπου μετά την ε, χρηματοδότηση παγκοσμίω 23 θα χρειαστεί να διαχειριστούμε φούσκες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό εδώ να μην επεκτείνουμε υπερβολικά τη χρηματοπιστωτική αγορά και να μην σκοτώσουμε την πίστοση γιατί είναι η μοναδική λύση που θα δώσει μια ανάσα στην πραγματική οικονομία. Θα πρέπει να δούμε επίσης και πιο αυστηρές απαιτήσει όσον αφορά τα παράγωγα και τα εσωτερικά μοντέλα λειτουργίας των τραπεζών. Συμφωνούμε με τις συγκεκριμένε ε, προτάσεις που αφορούν την πίστη, όπως επίσης και το εθνικό χρέος, όπως είχαμε και την ε, πρόσφατη ανακοίνωση το Σαββατοκύριακο για την Βασιλεία που αναφέρει κάτι σχετικά. Συμφωνώ λοιπόν για το 5-7 για το τραπεζικό κίνδυνο τραπεζών όσον αφορά το χρέος, το εθνικό χρέος. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τεράστιους κίνδυνους για τις ε, τράπεζες, γιατί έχουμε τον κίνδυνο πάντοτε του bail που θα εμπλέξει βέβαια τους ε, αποταμιευτές και θα έχουμε ολέθρες καταστάσεις σε κάποιες χώρες. Μετά, για τις επιπτώσεις των μη εξυπηρετωμένων δανείων, τα MPL. Δεν θέλουμε να βοηθήσουμε τα, αυτά τα funds που αγοράζουν πολύ χαμηλά τα δάνεια στο 10-15% και ξέρουμε ότι στην ουσία αυτοί είναι 4-5 ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι τέλο πάντων θα έχουν τεράστια κέρδη. Εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το πώ θα εφαρμοστεί. Είναι όμω πολύ σημαντικό οι τράπεζε να μην έχουν ζημιέ μεγάλε και που δεν θα είναι βιώσιμε μετά. Ε, συντάξεις, μισθή, οι κεφαλακές απαιτήσει. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία όσον αφορά τους ε, μικρομεσαίους οι οποίοι θέλουν να έχουν μια επιχειρήση, ένα σπίτι κτλ. Για τις υποδομές θα μπορούσαμε να μειώσουμε τις απαιτήσει, αλλά θέλουμε να υπάρχουν δομές με ενεργειακή απόδοση πραγματική ουσιώδη, απτή. Δεν θέλουμε μέσω τραπεζικού συστήματο να, να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τον άρθρακα και νομίζω ότι και εδώ οι πράσινοι συμφωνούν απόλυτα σε αυτό. Τέλος, ένα τελευταίο σημείο για, τις, για τους μισθούς. Νομίζω ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε πλήρως τους κανόνε που αφορούν τους μισθού των διοικητικών στελεχών και τα μπόνους. Ελπίζω οι συναντήσεις που θα υπάρξουν να είναι καρποφόρες, ιδιαίτερα μετά, το, μετά τις διακοπές και ελπίζω να έχουμε στο Κοινοβούλιο μια βιώσιμη πρόταση. Θα δούμε βέβαια στην πράξη τι θα προκύψει από την διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας, κατά 8 λεπτά διερμηνίας, πρέπει να ολοκληρώνουμε. Προβάνς Περές, Κάτσι 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μετά από τρεις ώρες που είμαι εδώ είναι καλό ε, που με επιτρέπει να μιλήσω τουλάχιστον 1,5 λεπτό. Ε, στα γαλλικά αφού βλέπω ότι η διερμηνής είναι εδώ. Να σας πω ότι το σημείο κίνησης αυτής της νομοθεσίας είναι οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών, ε, διαφορές μεταξύ των καθεστώτων των κρατών μελών. Βεβαίω έχει σημειωθεί πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. στα θέματα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωση. και όλα αυτά αλλάζουν το τοπίο μέσα στο οποίο εντάσσονται τα εθνικά συστήματα και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής εντάσσεται και στην διεθνή διαπραγμάτευση και πρέπει να δούμε πώς υπάρχει αυτός ο συσχετισμός και τι γίνεται με αυτόν. Με ξέπληξε όταν έμαθα ότι λέγεται ότι στο G20 σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια και τις ασφάλειες υπήρξε συμφωνία να μην έχουμε πια ανάλυση κινδύνων και αναλογικότητα κινδύνων βάσει μεγέθους του ε, τραπεζικού Ιδρύματος, αλλά βάσει της φύσης των στοιχείων ενεργητικών του εκάστοτε Ιδρύματος. Και θεωρώ ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις στο τραπεζικό τομέα και θα είναι αναπόδραστο. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, να μην το λάβουμε υπόψη μας. Είμαστε νομοθέτες, θα... ξέρουμε ότι θα έρθει και πρέπει να το προβλέψουμε. Όταν όμω το προβλέπουμε, αναλαμβάνουμε τον κινδύνο να εκθέσουμε τα δικά μας χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε επιπρόσθετους κινδύνους σε σχέση με τον ανταγωνισμό τους και πρόκειται δηλαδή για ένα εγχείρημα τετραγωνισμού του κύκλου. Εξού και είναι πολύ δύσκολο το καθήκον σας αγαπητές κύριε Σάιμον. Αλλά από εκεί και πέρα να σας πω τα εξή. Είπα δύο λόγια για την αναλογικότητα. Δεν μπορούμε να πούμε, όπως λέει ότι ο Σφεν Κίγκολτ, ότι δεν θέλουμε πια εθνική επιλογή και να έχουμε αναλογικότητα τελικά που θα οδηγήσει να έχουμε τελείως διαφορετικά ε, εθνικά συστήματα δεδομένης διαφορετικής αρχιτεκτονικής δομής του τροπεζικού συστήματος σε κάθε χώρα. Ε, ως προς τις πράσινες υποδομές και τις αποδοχές, να βρούμε μια κοινή γλώσσα και σε αυτά δεν αποτελεί μέρος της αρχικής πρότασης της Κομισιόν, αλλά είναι προτάσεις πολύ χρήσιμες, αγαπητοί κύριοι συγητά, και πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτές. Και αφού δεν έχω χρόνο, να διατρέξω την πλούσια πρόταση που μας κάνατε, θα μιλήσω μόνο για τον κίνδυνο των αγορών, το γεγονός ότι προετοιμάζεται νομοθεσία, υπάρχει από τη μία, επομένως θα ήταν αντιπαραγωγικό και αδέξιο οι Ευρωπαίοι να προδικάσουν εφαρμογή προτύπων που δεν έχουν οριστικοποιηθεί, ούτε αποφασιστεί, ούτε εγκριθεί ακόμα, ούτε ψηφιστεί και θα πρέπει να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα περαιτέρω. Ευχαριστώ όμως για αυτή τη βάση εργασίας και σίγουρα αυτό μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει και πολλή δουλειά, πολλή εργασία να γίνει. Επόμενη ομιλήτρια και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για, αυτό το, για αυτή τη δουλειά που έχει κάνει, πολύ σημαντική, και να κάνω και τέσσερις παρατηρήσεις πολύ γρήγορες. Σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις για θέματα κεφαλαϊκής επάρκειας και ρευστότητας για τις θηγατρικές, τις διασυνοριακές των τραπεζικών ιδρυμάτων. Μπορούμε να σημειώσουμε περισσότερη πρόοδο, να ε, μην αντιταχθούμε στην ανάπτυξη των διασυνοριακών τραπεζικών δραστηριοτήτων εντός Τραπεζικής Ένωσης, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα για την αναλογικότητα. Να επικεντρωθούμε στο reporting, στην υποβολή εκθέσεων, να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε η αναλογικότητα να μην οδηγήσει τελικά σε κατακαιρματισμό στην πράξη και ό,τι έχει να κάνει με την εφαρμογή των προτύπων της Βασιλείας να μην εσωματώσουμε υπερβολικά όλα αυτά που προβλέπονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην καταστούν οι δικές μας ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκές τράπεζες μη Ανταγωνιστικέ και μιλάω για τη συνολική ικανότητα απορρόφηση ζημιών, για την αναθεώρηση χαρτοφυλακίου συναλλαγών, ε, για το δίκτυο καθαρή σταθερή χρηματοδότηση και το ε, ε, όπως και οι συνάδελφος, ε, και εγώ συμφωνώ να μην βιαστούμε. Και η ίδια η Επιτροπή της Βασιλείας την επόμενη εβδομάδα είπε από μόνη της ότι θα τα ξαναδουλέψει αυτά τα στοιχεία. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν έχουμε άλλη διερμηνία. Ο κύριος Σίμων, παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι γεγονός. Σε μια άλλη συνεδρία θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Σίμων, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι πολύ σύντομος. Προς τον συνάδελφο Γκίγκολ δύο λόγια Χρειάστηκε πολύς χρόνος ε, για, ακριβώς για το λόγο που είδατε ε, ότι συζητήθηκαν και διάφορα επιχειρήματα σήμερα. Υπάρχουν κάποια θέματα που είναι καινούρια και θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε προς ποια κατεύθυνση ε, πρέπει να κινηθούμε και θέλουμε να βρούμε μια επικοδομητική λύση. Χαίρομαι που βλέπω ότι σε πολλά σημεία Ήδη υπάρχει κάποια συμφωνία και όταν θα έχουμε τις τροπολογίες θα μπορούμε να τις συγκεντρώσουμε και να προσπαθήσουμε τις τροπολογίες να τις συνενώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή λύση στην Επιτροπή. Για κάποια τώρα θέματα που, αφορά, που αφορούν το περιεχόμενο και ο συνάδελφος Κάρας ε, ε, έκανε κάποιες παρατηρήσεις. Όντως υπάρχουν ε, διάφορα θέματα για την, τους κινδύνους για το κλίμα, για τις πράσινες πράσινα περιουσιακά στοιχεία, κοινωνικές επιχειρήσεις. Εδώ έχουμε κάποιες διαφορές. Προσπαθούμε να δούμε αν όντω υπάρχει μικρότερος κίνδυνος. Ε, ε, ένα πολιτικό μήνυμα που δίνουμε και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν κάποια επιχειρήματα πολιτικού χαρακτήρα. Θέλουμε να ευνοήσουμε κάποιους τομείς της οικονομίας. θα είναι πιο ευνοϊκές οι πιστώσεις για ε, κάποιους τομείς της οικονομίας. και για την κινητικότητα που θέλουμε να ενθαρρύνουμε. Όταν θέλουμε να ενθαρρύνουμε κάποιους τομείς, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δώσουμε τα σχετικά κίνητρα. όταν δίνονται salary backed loans, μια ιδέα που ξεκινάει από την Ιταλία. Δίνεται ένα είδος εγγύησης, ούτως ώστε η τράπεζα να μην έχει κίνδυνο και ο πελάτης έχει πολύ καλά επιτόκια για την πίστοση που παίρνει. Η χορήγηση τέτοιων ε, πιστώσεων μπορεί να είναι μια λύση την οποία θα επιλέξουμε. Δεν θέλω να κάνω τις ε, παρατηρήσεις για όλα τα σχόλια σήμερα, αλλά σίγουρα θα μας δοθεί ευκαιρία να τα συζητήσουμε και στην Επιτροπή Οίκων, αλλά και σε συζητήσεις με τους συναδέλφους. και ελπίζω ότι θα προλάβουμε εγκαίρως να κλείσουμε το φάκελο αυτό. Και ευχαριστώ βέβαια και τους σκιώδεις συζητητές για την εξαιρετική συνεργασία μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ και τους διερμηνείς, λέει ο που δείχνουν ευελιξία και έμειναν περισσότερο. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 25 Ιανουαρίου. για την ε, CRD και 24 Ιανουαρίου για ε, το CMR. 21 και 22 Φεβρουαρίου θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα λοιπόν και θα τα πούμε μετά τα Χριστούγεννα.